Okay, let's start, dear colleagues. I sub, I submit... Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σα υποβάλλω προ έγκριση τις εξή αλλαγέ. Θα αναβληθεί η ψηφοφορία από τι 15 ε, Σεπτεμβρίου. Η κοινή ακρόαση στι 15 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει μέχρι τη μία η ώρα στην αίθουσα Jam 2Q, το σημείο 26 για τι στρατηγικέ αιτήσεις του όρομα 2015 θα αναβληθεί για την επόμενη συνεδρία τη ΛΥΠΕ, τα σημεία 27-29 για την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων σε σχέση με τα πλουροσκοπικά δεδομένα στη Σουηδία, του Βαλτίο και στην Πολωνία θα ξεκινήσει στι 5 παρα 10, το σημείο 30 για το VIS, η παρουσίαση του σχεδίου έκθεση. έχει προσθεθεί στην παρουσίαση του Συμβουλίου και θα ξεκινήσει στις 5 σημείο 31 για τη Συμφωνία Ομπρέλα Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ θα παρουσιαστεί από τις 5.25 μέχρι τις 6. Και μια έκτακτη συνεδρίαση των συντονιστών θα ξεκινήσει από τι 6 και μετά για κλεισμένο των θυρών. Αν δεν υπάρχουν θα εγκρίνεται με τη διάταξη όπως τροποποιήθηκε. να σας ενημερώσω ότι δεν έχουμε δυστυχώ διερμηνία στα κρατικά και στα ελληνικά σημερινή συνεδρίαση. Και τώρα θα περάσουμε στην έγκριση των ε, συστάσεων των συντονιστών. Ιρκόφ, ECR Ο κύριος ε, Κύρκοπ είναι εδώ και έχει διοριστεί ως εισηγητής ε, πρόσβαση για την διαβούλευση του ΒΙΣ από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και από την για τους σκοπούς της πρόληψης, ε, έρευνας ε, των τρομοκρατικών υποθέσεων και άλλων σοβαρών πενικών αδικημάτων. Η κυρία Φλασικό Φλασσικό-Βαμπένοβα έχει διοριστεί ως εισηγήτρια για τις τρεις ακόλουθες εκθέσεις για την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων σε σχέση με τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σουηδία, την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων σε σχέση με τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στο Βέλγιο και αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων σε σχέση με τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Πολωνία. Ε, ο κατάλογος ε, των συστάσεων των συντονιστών συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα. Εγκρίνει η Επιτροπή της συστάσεις αυτές από τους συντονιστές. Ωραία, σας ευχαριστώ. Εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 8ης Ιανουαρίου 5 Φεβρουαρίου και 24 Φεβρουαρίου και 26 Φεβρουαρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Περνάμε τώρα στα σημεία 4, 5, 6 και 7. Τα επόμενα σημεία στην ημερησία διάταξη αφορούν παρουσιάσει από το Συμβούλιο και τι Κομισιόν και την εξέταση των σχεδίων εκθέσεων για τέσσερι μη νομοθετικέ προτάσει για την υποβολή νέων ψυχοτρόπων ουσιών σε μέτρα ελέγχου. Η προθεσμία των ε, τριών μηνών για διαβούλευση ξεκινά την ημέρα μετά την λήψη της επιστολής στο Κοινοβούλιο, δηλαδή ολοκληρώνεται την 7η Οκτωβρίου. Επειδή πήγε το θέμα, οι συντονιστέ ΛΥΜΠΕ αποφάσισαν στη συνεδρία στι 7 Σεπτεμβρίου να εργαστούν μόνο στα αγγλικά. Τώρα, θα δώσω το λόγο στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν για να παρουσιάσουν και τις τέσσερις προτάσεις και κατόπιν ε, στους εισηγητές. Ο κύριος Ματιέ Κόνερ, εκ μέρους της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 16 ε, Απριλίου 2015 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι θα πρέπει να διαβουλευτούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πριν να υιοθετήσουμε μία νέα απόφαση για να υποβάλουμε νέες ψυχοτρόπες ουσίες ε, στην απόφαση ε, που προβλέπεται 2005-86 για να σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου και να λάβουμε υπόψη την νέα διαδικασία που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο. Η Ριζόντια ομάδα για τα ναρκωτικά έχει αναθεωρήσει τώρα τι αρκές προτάσεις της Κομισιόν. Ε, έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή εκτελεστικέ αποφάσει, το σχέδιο των εκτελεστικών αποφάσεων που υιοθετούν από το Συμβούλιο. Ο στόχο αυτών των τεσσάρων εφαρμοστικών αποφάσεων είναι να επιβληθούν σε μέτρα ελέγχου μια σειρά νέων επικίνδυνων ψυχοτρόπων ουσιών και ε, ουσιαστικά πρόκειται για νόμιμε ουσίε που είναι προσβάσιμε σε χρήστε και ουσιαστικά αποτελούν ε, εναλλακτικέ ουσίε για την κατανάλωση ναρκωτικών Επίσης, οι κίνδυνοι είναι συχνά ε, μη γνωστοί και ε, ουσιαστικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με προσπάθειες καταπολέμησης της ε, τοξικομανίας. Οι προτάσεις που έχουμε υποβάλει θα χρησιμοποιήσω τώρα τα σύντομα ονόματα γιατί είναι πολύπλοκα ολόκληρες οι ονομασίες. Σε ό,τι αφορά τις ψυχότροπες ουσίες, έχουμε τέσσερα φετιναφημενημένοι είχαμε ε, θανάτους στα κράτη-μέλη. Η δεύτερη νέα ψυχοτρόπος ουσίας είναι η 5-2 αμυλπροπενδολίου και έχουν αναφερθεί τέσσερις θάνατοι σε τέσσερα κράτη-μέλη και πάλι δεν υπάρχει γνωστή ιατρική χρήση. Οι νέες ουσίες που αφορούν την τρίτη απόφαση εφαρμογής και που πρέπει να βάλουμε υπό έλεγχο, δηλαδή το 25 INBOM, και την ε, AH7921 και το MDPV επίσης έχουν συνδεθεί με πολυαριθμούς θανάτους στην Ένωση ε, και είχαμε 180 ε, θανάτους που έχουν συνδεθεί μόνο με το MDPV και έχουν αναφερθεί από 8 κράτη-μέλη τουλάχιστον και σε ό,τι αφορά την τέταρτη ψυχοτροποσία που θα υποβληθεί σε μέτρα ελέγχου ε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ουσία 4,4 DMAR έχει συνδεθεί τουλάχιστον με 31 θανάτους σε τρία κρατημέλη και η άλλη ουσία, η MT45, έχει συνδεθεί με 28 θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τονίσω ότι για όλες τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες που θα επιβληθούν σε μέτρα ελέγχου δυνάμει των σχεδίων αποφάσεων, ε, οι επιπτώσεις για τη δημόσια και την ατομική υγεία θα είναι σημαντικές ε, αν ε, οι ουσίες αυτές διαδοθούν περισσότερο. Τα στοιχεία που έχουμε από τις εκθέσεις του παρατηρητηρίου μας δίνουν επαρκείς λόγους για να θέσουμε αυτές τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες σε μέτρα ελέγχου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου του 2005. Η Προεδρία του Συμβουλίου πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την άποψη ότι οι παραπάνω ψυχοτρόπε ουσίε θα πρέπει να υποβληθούν σε μέτρα ελέγχου έτσι ώστε τα εφαρμοστικά μέτρα, τα εκτελεστικά μέτρα να μπορούν να υιοθετηθούν σήμερα το συντομότερο δυνατό. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κυρία Μετά. Εκ μέρους Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, λίγα πράγματα έχω να προσθέσω στα ως επιπροεδρία. Να θυμίσω γιατί προτείναμε να απαγορεύσουμε αυτές τις οκτώ ουσίες που συζητούμε σήμερα. Οι νέες αυτές ουσίες ανέκαθεν συνδέονταν με θανάτους και δηλητηριάσεις είναι πολύ βλαβερές, αντιπροσωπεύουν κίνδυνο εξάπλωσης ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές περιπτώσεις πολλούνται ως εναλλακτικές λύσεις υποκαθιστώντας παράνομες ναρκωτικές ουσίες. Πολλές φορές πολλούνται και μέσω διαδικτύου. Καμία από αυτές τις ουσίες δεν έχει καθιερωμένη ιατρική χρήση. Τέσσερις προτάσεις υποβάλαμε εκ των υστέρων μετά από την απόφαση 37 2005 του Συμβουλίου για τέσσερις λοιπόν επιπλέον ουσίες. Η Επιθυμονική Επιτροπή εκπώνησε πόρισμα βάσει του οποίου η Κομισιόν θεωρούσε και θεωρεί ότι υπάρχει πλέον λόγος ευρεία απαγόρευση αυτών των ουσιών κατά κύριο λόγο διότι είναι βλαβερέ και δεύτερο διότι προσωμιώνουν τα αποτελέσματα τη επιπτώση απαγορευμένων ουσιών. Αποτελούν λοιπόν αυτέ οι ουσίε κίνδυνο και γι' αυτό θεωρούμε ω Κομισιόν ότι πρέπει να δράσουμε αμέσω. Ευχαριστώ. Πρώτο ευχαριστώ. Κύριε Πόνι, εισηγητή των τεσσάρων εκθέσεων 2013-2021 ε και 2014 0304 αλήθεια το λόγο Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι να σας παρουσιάσω εν συντομία δύο εκθέσεις επί του σχεδίου εφαρμοκτικής απόφασης του Συμβουλίου έχουμε τρεις εδώ ψυχοτρόπους ουσίες που πρέπει να υποβληθούν σε μέτρα ελέγχου και στις δύο περιπτώσεις έχουμε δύο αποφάσεις που προαναφέραμε του Συμβουλίου. Η πρώτη υπαριθμών 2014 κάθετος 340 αφορά υποβολή σε μέτρα ελέγχου την Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο ουσίες. Θα τις αναφέρουμε με την κοινή του ονομασία 4, 4 DMR και MT 45. Και οι δύο αυτές ουσίες αξιολογήθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού για την Πρόληψη των Ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθησαν τα σχετικά πορίσματα στις 19 Σεπτεμβρίου του 2014 κοινοποιήθηκε η ουσία στο σύστημα εγγύησης Προδοποίηση τον Δεκέμβριο του 2012. 31 θάνατοι σημειώθηκαν σε πολλές χώρες μεταξύ του Ιουνίου του 2013 και του Ιουνίου του 2014. Δεν έχει προκύψει όμως καθιερωμένη ιατρική ή κτηνιατρική ή άλλη χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των ουσιών. Οι ουσίες αυτές, εκ των οποίων η πρώτη λέγεται MT45, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ουσία, η έκθεση υπευλήθη σε Επιτροπή και Συμβούλιο 6 Οκτωβρίου 2014. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, 28 θάνατοι είχαν καταγραφεί μεταξύ του Νοεμβρίου του 2013 και του Ιουλίου του 2014. Ούτε αυτή η ουσία έχει γνωστή ιατρική, την ιατρική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο ουσίες δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση του ΟΗΕ σχετικά με την, τον έλεγχο των ναρκωτικών ουσιών, ούτε περιλαμβάνονται στην σύμβαση για, του ΟΗΕ πάντα για τις ψυχοτρόπους ουσίες. Δεν είναι αξιολόγηση, ούτε θα αξιολογηθούν από ό,τι φαίνεται στο πρόσχες μέλλον από τον ΟΗΕ. Γι' αυτό έχουμε κάθε λόγο να προβούμε εμεί σε ρύθμιση ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο ουσίες έχει αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνε σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή και συντρέχουν όλοι οι λόγοι και προϋποθέσεις για να προβούμε στη λήψη μέτρων. Προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε την απόφαση του Συμβουλίου. Το ερώτημα είναι γιατί καθυστερήσαμε τόσο, γιατί αλλά με δράσει τώρα μόλις, ενώ έχει περάσει τόσο χρόνος από τη στιγμή που γνωρίσαμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των ουσιών. Θέλω να θυμίσω προκειμένου ότι εργαζόμαστε στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος που επιτρέπει πλέον προσωρινές απαγορεύσεις. Δηλαδή οι ουσίες μπορούν να απαγορευτούν έστω και προσωπικά από τη στιγμή της πρώτης έστω και προκαταρκτικής ανάλυσης. Απαγορεύεται λοιπόν η κυκλοφορία τους στην ε, αγορά, αλλά χρειάζεται να περιμένουμε ένα χρόνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπερψηφίσει τη θέση του τον Απρίλιο του 2014, όμως το Συμβούλιο ακόμη την επεξεργάζεται χωρίς να έχει καταλήξει απόφαση. Γι' αυτό και καλό την Προεδρία του Λουξεμβούργου να επιταχύνει τις σχετικές εργασίες. Το πρόβλημα όμως οξύνεται, αυτό το γνωρίζουμε. Όλο και περισσότερες νέες ουσίες εφευρίσκονται και δυστυχώς τα θύματα αυξάνονται και αυτά. Η Ευρώπη δεν έχει εργαλεία για άμεση δράση κατά αυτών των ψυχοτρόπων ουσιών, των ενεργών ψυχοτρόπων ουσιών. Ας μην χάνουμε λοιπόν χρόνο. Η δεύτερη έκθεση που θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα αφορά το σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης του Συμβουλίου για την άλλη ουσία, την αμφεταμίνη 2013-0021 διαδικασία διαβούλευσης. Η εκτίμηση, η αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα εφήγης για την Κομισιόν στις 29 Νοεμβρίου του 2012. Η εν ουσία έχει ανοιχνευθεί σε 15 κράτη-μέλη. Καταγράφηκαν σε 21 θάνατοι. Η ουσία είναι ακροστοξική και τα στοιχεία δείχνουν υψηλότερο κίνδυνο όταν ε, συνδέεται η λήψη της με τη λήψη άλλων ουσιών. Δεν έχει καταγεγραμμένη η γνωστή ιατρική ή κτηνιατρική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και άλλες δύο ουσίες δεν αξιολογείται από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Συνεπώς, οφείλουμε να αναλάβουμε δράση. Η απόφαση αυτή υποκαθιστά την απόφαση του Συμβουλίου 29 του 2013 που ακυρώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Απριλίου του 2015. Το κύριο αποτέλεσμα από αυτήν την απόφαση είναι ότι το Συμβούλιο οφείλει να διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν λαμβάνει σχετικέ αποφάσει, κάθε φορά δηλαδή που υποβάλλονται ενεργέ ψυχοτρόποι ουσίε εν ώψη λήψη μέτρων, κάτι το οποίο συμβαίνει σήμερα. το καθεστώς αυτό θα συνεχίσει να ισχύει ως ότου φυσικά αντικατασταθεί από το νέο. Προτείνω την υπερψήφιση του σχεδίου της απόφασης έτσι ώστε η ουσία αυτή και αυτή η ουσία να παραμείνει αντικείμενο μέτρων ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ για την υπερψήφιση και ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν και το Συμβούλιο για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ. Βάριο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο αλλά και την Κομισιόν και τον κύριο Μπον για την παρέμβασή του και για την εργασία του. Εγώ δεν θα επαναλάβω το πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο σε σχέση με την ανείχνευση νέων ψυχοτρόπων ουσιών. Σήμερα παρουσιάζω δύο εκθέσεις. Ε, δεν ε, έχει κατατεθεί καμία τροπολογία στην πρόταση του Συμβουλίου το μήνυμα είναι σαφέ, πρέπει να αποβληθούν αυτές οι ουσίες σε μέτρα ελέγχου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο και να υπάρχει διασυνοριακή δικαστική συνεργασία και προστασία των καταναλωτών κατά των κινδύνων που μπορεί να θέσει η κατανάλωση αυτών των ουσιών. Η πρώτη έκθεση που παρουσιάζω, γιατί έχουμε δύο όπως σας είπα, έχει να κάνει με την ε, ουσία που λέγεται 25-INBOME. Η δεύτερη ε, ουσία είναι η AH7921. Η τρίτη ουσία είναι η MDPV. Σε τρία κράτη-μέλη έχουν καταγραφεί τέσσερις συναφείς θάνατοι με την 25 INBOME. Σε τέσσερα κράτη-μέλη ε, είχαμε σοβαρή τοξικότητα ε, με την κατανάλωση και με την κοινοποίηση 32 περιπτώσεων δηλητηρίαση, μη θανατηφόρου. Ε, αυτή η κατανάλωση των νέων ουσιών, αν αυξηθεί, οι συνέπειες θα είναι σημαντικές για τη δημόσια υγεία. 22 κράτη και η Νορβηγία κοινοποίησαν ε, στο ε, Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης της Ταξικομενίας ε, ότι υπήρχε στα 25 κράτη η παρουσία της ουσίας 25ANOME σύμφωνα με τους καταναλωτές, οι παρενέργειες της AH7921 μοιάζουν με κλασικά οπιοειδή και προκαλούν ε, μια εφορία. Η MDPV ε, ουσιαστικά έχει ένα προφίλ ανάλογο της μεθαμφεταμίνης και της κοκαίνης, αν και μπορεί να διαρκεί περισσότερο. Τον ε, Σεπτέμβριο του 2009 και τον Αύγουστο του 2013 είχαμε θανάτους σε 8 κράτη-μέλη. Δεύτερη έκθεση αναφέρεται ε, στην ουσία 5-2 ενδόλιο. Η τοξικότητα τοξικότητα, η οξία τοξικότητα της ουσίας αυτής μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο παρενέργειες όπως υποθερμία, ταχυκαρδία, μυδρίαση, τρέμουλο κοινοποιήθηκε στο κέντρο παρακολούθησης της τοξικομανίας και της Europol ότι ενηχνεύτηκε η ουσία ΑΣΥ. Καθώς αυτές οι ουσίες θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία των πολιτών, ζητώ την υποστήριξη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για να μπορεί το Συμβούλιο να θέσει σε μέτρα ελέγχου αυτές τις ουσίες. 27 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία και η ψηφοφορία στην Λίμπε θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να εκφράσω μια μεγάλη ανησυχία, όπως και ο κύριος Μπόνη, για τη σημερινή κατάσταση του κανονισμού και της οδηγίας σχετικά με τις νέες ψυχότροπες ουσίες που εγκρίναμε πέρσι στο Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε επιγόντως ένα σύστημα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ένα μηχανισμό που να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε νέες ψυχοτρόπες ουσίες, οι νέες επικίνδυνες ουσίες να απαγορευτούν πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα. Ζητώ από το Συμβουλίο να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών για να πετύχει μια καλή συμφωνία επί της νομικής βάσης των δύο νομοθετημάτων. Και δεν το ζητώ μόνο εγώ, αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έτσι ώστε νέες επικίνδυνες ουσίες να απαγορευτούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προϊόν κατανάλωσης. Σας ευχαριστώ. Thank you. Now it's time for... Ευχαριστώ. Οι σιώδεις εισηγητές έχουν τώρα το λόγο. Όποιος θέλει βεβαίως να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν. Ενδεχομένως η Επιτροπή, το Συμβούλιο. Α, κύριε Στίβενς. Η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την εξαιρετική παρουσίαση και για το σχέδιο κειμένου που συζητούμε σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχω κάποια σχόλια να κάνω, αλλά όχι πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να συνεχίσουμε αυτή την συνεργασία και στο μέλλον. Οι τροπολογίες για τις 17 Σεπτεμβρίου μόνο στα αγγλικά στις 12 θα εξεταστούν στις 22 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και τον Οκτώβριο 5 με 8, το αργότερο δηλαδή 7 Οκτωβρίου θα πρέπει να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Δεν βλέπω να ξαναθέλετε το λόγο. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο σημείο αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η παρουσίαση της ε, έκθεσης από τον κύριο Γκάμπριελ. Πρόκειται για το θέμα των θεωρήσεων και αλλαγή υποχρέωσης ε, από μέρους 9 ετών. Βεβαίως όσον αφορά τα ελεύθερα, την ελεύθερη μετακίνηση για τους ε, πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις εννέα χώρες οι οποίες για 90 ημέρες επιτρέπουν αυτήν την διαμονή Το τέλος της επεξεργασίας του κειμένου έγινε στο τέλος του 2014, κατόπιν το Μάιο του 2015 ψηφίστηκε, αυτές οι συμφωνίες ε, έχουν πάει στο Συμβούλιο. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Γκάμπριελ, τον εισηγητή, και κατόπιν στους κυρία. Απαλλαγή και κάπως αλλιώς το λένε. Άρση, άρση Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία μου. Θα παρουσιάσω τις εννέα θέσεις που αφορούν αυτήν την απαλλαγή υποχρέωση θεώρησης για τις χώρες αυτές, τις εννέα χώρες, ε, την τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Τρινιντάδ και οι υπόλοιπες χώρες, η νήσι Σαμόα. Πρόκειται για τις ε, υπογραφές αυτών των ε, συμφωνιών που έγιναν μετά από τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κάθε μία από αυτές τις χώρες, οι οποίες ήδη αυτές οι απαλλαγές έχουν αρχίσει να ισχύουν προσωρινά. Και τώρα περνάμε στην μόνιμη φάση, στην τελική φάση αυτών των συμφωνιών. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροπολογιών, θα πρέπει δηλαδή απλώς να τις δεχτούμε ή να τις απορρίψουμε ε, ξεχωριστά την κάθε συμφωνία. Πέρα λοιπόν από την διαδικασία μπορώ εδώ να σας ε, επισημάνω κάποια συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, όσον αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεύτερον, ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την απαλλαγή των ε, υποχρεώσεων θεώρησης. Θέλησα να παρουσιάσω την συμβολική αλλά και την πολιτική αξία αυτών των συμφωνιών με τις εννέα αυτές χώρες. Πρόκειται για έναν τρόπο να εντετικοποιήσουμε αυτόν τον πολιτικό διάλογο, ιδιαίτερα για θέματα θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραδείγματο χάρη για τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήδη μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια τεχνική ομάδα εργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, Εμμυράτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως μετά τη σύναψη αυτής της συμβολίας θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον πολιτικό μας διάλογο με τις χώρες ΑΚΕ για θέματα όπως τη θανατή και την ισότητα ανδρών και γυναικών. Δεύτερον, αυτές οι συμφωνίες δίνουν κάποιες οικονομικές δυνατότητες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις τρίτες χώρες όσον αφορά την αύξηση των τουριστικών ροών, τη βελτίωση των οικονομικών αλλά και τουριστικών συναλλαγών και επενδύσεων. Για όλες αυτές τις χώρες τα ποσοστά άρνησης ε, θεωρήσεων ιδιαίτερα για ε, διαμονές μικρής διάρκειας και τουριστικές επισκέψεις είναι εξαιρετικά χαμηλές. Όπως βλέπουμε, οι περισσότερες αιτήσει γίνονται δεκτές, όπως παραδείγματο χάρη για χώρες όπως το Τρινιτάτ και το Μπάγκο και βλέπουμε ότι οι περισσότερες αυτών των αιτήσεων γίνονται δεκτές και ότι υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη. Για τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ θα ήθελα να πω ότι εμείς στα πλαίσια των συζητήσεών μας μπορούμε να κάνουμε μία σειρά παρατηρήσεων και σχολείων. Για άλλη μια φορά θα ήθελα εδώ να ακούσουμε από μέρους της Επιτροπής κάποιες λίγο πιο ικανοποιητικές απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Πρώτον, όσον αφορά την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την παρακολούθηση και την πρόοδο αυτών των διμερών συμφωνιών, ιδιαίτερα μέσω των μεικτών επιτροπών διαχείρισης αυτών των συμφωνιών. Μια απάντηση που περιμένουμε από την Επιτροπή στην γραπτή ερώτηση που είχαμε θέσει για τα σημεία αυτά. Μετά λοιπόν την θέση σε ισχύ της συμφωνίας θα πρέπει να τηρούνται τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο κείμενο της συμφωνίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την αμοιβαιότητα αλλά και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να υπάρχει πραγματική αμοιβαιότητα όσον αφορά τη μεταχείριση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχέτως από ποια χώρα προέρχονται. Η προσωρινή θέση σε ισχύ της συμφωνίας πριν την έγκριση της Ευρωπαϊκής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούμε ότι θέτει σε κίνδυνο την ε, συμφωνία και την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είχαμε πει ότι οι συμφωνίες αυτές μπορούν με μεγάλη ταχύτητα να υλοποιηθούν από τη στιγμή βεβαίως που θα μπορέσει να γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμμετάσχει σε αυτήν την διαδικασία. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, του συναδέλφους, ιδιαίτερα τους και συζητητές για τη συνεισφορά τους σε αυτή την εργασία. Και ολοκληρώνω ζητώντας σας ε, να στηρίξετε αυτήν την συμφωνία υιοθετώντα της προς όφελος των πολιτών των εννέα αυτών χωρών αλλά και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα σκιώδεις, εισηγητές. Α, η Επιτροπή. Πρώτα η Κομισιόν παρακαλώ. Ποιο θέλει πρώτα στο λόγο, Συμβούλιο, Κομισιόν ή Κομισιόν. Κυρία Πρόεδρε, μόλις έφτασα δυστυχώς, δεν γνωρίζω τι διημήρθη, τι είπε η κυρία Γκάμπριελ, τι δημιουργήθηκε τι διάβασα βέβαια στην εκθεσή της και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί βεβαίω είναι θετική η σύσταση. Προσβλέπουμε στην λήψη της ε, σύμφωνης του Κοινοβουλίου για αυτές τις συμφωνίες. Γνωρίζω, έκανε μια παρατήρηση για το θέμα της εφαρμογής από την ημέρα της υπογραφής. Επ' αυτού να πω ότι ακολουθούμε απλώς το προηγούμενο, ότι κάναμε δηλαδή σε παρομοίες συμφωνίες εξαίρεσης. Το 2009, για παράδειγμα, ενημερώσαμε και ενημερώνουμε την Επιτροπή με επιστολή του Γενικού μου Διευθυντή τον Μάρτιο του 2015. Ενημερώνουμε δηλαδή, έχουμε ενημερώσει από τον Μάρτιο του 2015 ότι οι εν λόγω συμφωνίες δεν σε ισχύ από την ημερομένη της υπογραφής τους. Είναι κάπως παράδοξο να δώσει τη σένεσή του το Κοινοβούλιο σε μια συμφωνία βεβαίως η οποία ήδη ισχύει. Παρ' όλα αυτά αυτό είναι το προηγούμενο. Και ξέρετε, δεν υπήρξαν αντιρρήσιτικά με τις συμφωνίες αυτές. Δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη συζήτηση, ούτε εκκρεμεί κάποιο ζήτημα που θέλει περαιτέρω συζήτηση. Εννοείται ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη δώσει τη σύνδεση του για την μεταφορά αυτών των χώρων στον λεγόμενο θετικό κατάλογο. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ε, όλα αυτά τα στοιχεία, πιστεύω ότι η θέση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής δεν θα έπρεπε να θεωρείται ως δυσκολία. Αυτά. Ευχαριστώ κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ πολύ για την θερική σας σύσταση και την έκθεση. Θα τα ξαναπούμε βεβαίω γιατί εκκρεμούν και άλλες παρόμοιες συμφωνίες απαλλαγή από υποχρέωση θεώρησης που διαπραγματευθήκαμε στο ίδιο πλαίσιο. Άρα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε αργότερα φέτος το, εντός του 15 προεδρό. Ευχαριστώ. Δεν ζήτησε κανεί άλλο το λόγο. Από τους όμω, όμως. Όχι. έχουμε ένα. Ναι, κυρία Στιβένση. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω εκ νέου την εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα θετικό σήμα για περισσότερη επαφή με τους τοπικούς πληθυσμούς, για περισσότερες ευκαιρίες ταξιδιών, τουρισμού αλλά και επιχειρηματικών συνεργασιών. Οι συμφωνίες αυτές θα είναι θετικές για τους πολίτες των χωρών που ταξιδεύουν συχνά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα μπορούν να παίρνουν να διάρκεια για τα διάφορα ταξίδια τους. Σημείωσα επίσης το ότι δεν απειλείται ο χώρος Σέγγεν ε, όσον αφορά η λόγω αν θέλετε της παρανομής μετανάστευσης. Ειδικά όσον αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πραγματικά ελπίζουμε ότι η συμφωνία θα αποτελέσει και ένα επιπλέον κίνητρο και μέσο, μια δυνατότητα για να αντιμετωπίσουμε την δημοκρατία αλλά και τη μεταβολή του κλίματος. Επίσης, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυρά, θα θελήσουμε και προβλήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, ελευθερία έκφρασης καθώς και μετακινήσεων εργαζομένων. Προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία με όλους σας. Ευχαριστώ. Κύριε Κιλίμ. Συγγνώμη, και εγώ την τελευταία στιγμή έφτασα, αλλά θέλω να συγχαρώ και εγώ την Μαρία για την σκληρή της δουλειά. Μελέτησε το θέμα σε βάθος, δούλεψε πολύ συνεργάστηκε εξαιρετικά με τους ε, ισκιώδεις ηγητές, όπως πάντα το κάνει. Δεν έχω να πω κάτι για το ε, σχέδιο, με εξαίρεση δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ως προς τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που έθεσε η κυρία Στίβενς, να πω και εγώ ότι αυτός ο τύπος συμφωνίας. Πρώτον, διευκολύνει την κινητικότητα, την ανάπτυξη οικονομικών δεσμών, ε, αλλά και από την καθαρά ανθρώπινη σκοπιά στο ρημαίο τη επιστήμης και του πολιτισμού θα έχουμε περισσότερες ανταλλαγές, ε, θα έχουμε περισσότερες επαφές μεταξύ των δύο λαών. Όσον αφορά κάτι τελείως διαφορετικό, έχει μεγάλη σημασία το Κοινοβουλίο να παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των συμφωνιών. Διότι έχουμε καμιά φορά την εντύπωση ότι ωραία δίνουμε τη συνέντευξή μα και μετά σταματούν τα πάντα, ε, κανείς δεν μα ενημερώνει μετά. Και το λέω αυτό πολύ μάλλον καθώ. και είναι κάτι που έχουμε συζητήσει και ζητήσει πολλέ φορέ ε, ότι όπω έλεγα η παρέμβαση του Κοινοβουλίου επέρχεται ενώ ήδη ισχύουν, έχουν μάλλον τεθεί σε ισχύ οι συμφωνίες ε, κάτι που δεν έχει πολύ ενθαρρυντικό για μας βεβαίω, έστω και σε προσωρινή βάση. Να το δούμε αυτό. Και τονίζω επίση την δημιουργία μηχανισμού στη βάση της αμοιβαιότητας. Εν γέννη λοιπόν με υπέρ τη συμφωνίας, υπέρ των συμφωνιών. Όμω πρέπει, στην περίπτωση που για παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκφράσουν την επιθυμία να έρθουν λίγο πιο κοντά σε εμά. Μπορεί μάλλον να έχουν δείξει την θέλησή του να έρθουν πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, των γυναικών κλπ. Ε, στον τομέα τη ελευθερία τη έκφραση έχουν επικώ πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είμαι λοιπόν υπέρ τη συμφωνία, αλλά έχω και τι επιφυλάξει που μόλις ε, σας ε, ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκάμπριελ, αν το επιθυμεί, για να κάνει μία σύνοψη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους κοιόδες, την κυρία Στίβενσον για την ε, παρατήρησή της. Ευχαριστώ την Επιτροπή για κάποιες αρχές απαντήσεων που μας έδωσε. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει πραγματικά να δημιουργήσουμε προηγούμενα τα οποία να μπορούν να λειτουργήσουν στη διάρκεια του χρόνου. Ευχαριστώ και την Σκιώδη, την κυρία Γκυγιόμ. Πάντα πρέπει να ενημερωνόμαστε καλύτερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι εδώ για να θέτει εμπόδια για να εμποδίζει τη διαδικασία. Μπορούμε και εμείς να εργαστούμε με συνοπτικές διαδικασίες και γρήγορα, αλλά πάντα θα πρέπει να σεβόμαστε τις συνθήκες και να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως πρέπει. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι θέλουμε πληροφορίες όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες. 19 χώρες θα πρέπει να εξεταστούν και θα θέλαμε για χώρες όπως η Κολομβία παραδείγματο χάρη να μην βρεθούμε στην ίδια κατάσταση όπως αυτή που βρεθήκαμε με τις εννέα αυτές χώρες. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Επαναλαμβάνω ότι η συνεργασία μας ε, έχει ξεκινήσει με πολύ ικανοποιητικό τρόπο, θα πρέπει να λογιστεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, 21 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι και βεβαίως ότι θα γίνουν δεκτές μόνο διαδικαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. περιμένουμε. Σας περιμένουμε μάλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα περάσουμε στο θέμα του πακέτου που αφορά τις θεωρήσεις. Καταρχήν το θέμα του κώδικα θεωρήσεων και δάνω το λόγο στον κύριο Ακύλας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, για μια φορά είμαστε μπροστά στη διαχείριση του χρόνου στην Επιτροπή αυτή. Έφτασα ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για την παρουσίασή μου. Για να παρουσιάσω αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, σε σχέση με την διατύπωση του Ενωσιακού Κώδικα Θεωρήσεων. Εδώ και μήνες εργαζόμαστε επί αυτής ε, της αναδιατύπωσης ε, και αναφέρεται αυτό και στην θεώρηση περιοδίας Ρίνδικα που θα παρουσιαστεί σήμερα από κοινού με το πακέτο θεωρήσεων. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για το έργο της, για τη διαχείριση της έκθεσης αυτής, καθώς ε, και την Τάνια Φαγιών, τη συνάδελφο από την ομάδα μου η οποία με βοήθησε εν μέρη στην εκπόνηση αυτού του φακέλου, αλλά θα περάσω τώρα στην παρουσίαση της έκθεσης ε, ως ε, ένα αποτέλεσμα έντονης δουλειάς, όπου προσπαθήσαμε να βάλουμε ε, τις συνεισφορές των σκιωδών εισηγητών, αλλά και όλων των συναδέλφων που κατέθεσαν τροπολογίες. Στην παρουσίαση των γράφων εργασίας πριν λίγων μήνες και κατόπιν της ακρόασης που έλαβε χώρα. Εγώ όλο αυτό το καιρό είχα μία σειρά ε, συναντήσεων με κυβερνητικέ οργανώσεις, με ομάδες ε, συμφερόντων που ενδιαφέρονται για αυτή την νομοθετική πρόταση της Κομισιόν και είχα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και με ακαδημαϊκούς, με καθηγητές που ειδικεύονται στο ανθρωπιστικό δίκαιο και λόγω του αντικτύπου αυτής της νομοθεσίας ε, σε πολίτες τρίτων χωρών και έχοντας κατά νου ότι έχουμε εδώ μία νομοθεσία που εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη στα προξενικά δίκτυά τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας φάνηκε καλό να οργανώσουμε και μία διερευνητική αποστολή προξενία στο εξωτερικό για να αξιολογήσουμε πώς λειτουργεί στην πράξη το σύστημα των θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά αυτό θα μπορούσε να συμπληρώσει αυτό το σχέδιο. Και αυτό είναι πρώτο τώρα γενικό σχόλιο. Ήδη προχώρησε στην παρουσίαση του εγγράφου εργασίας η φιλοσοφία της πρότασης της Κομισιόν βασικά είναι κατάλληλη. Εδώ ο σκοπός είναι η διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων, επικαιροποιώντας τον ενωσιακό κώδικα θεωρήσεων για να διορθωθούν προβλήματα στη λειτουργία που έχουν εντοπιστεί με το πέρασμα του χρόνου και για να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό που έχει ο κώδικας θεωρήσεων ως προς την προώθηση ε, των ανθρώπινων ανταλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου. Φυσικά ο κόσμος ε, είναι όλο ένα και πιο αλληλεξαρτώμενος. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα πιο υψηλά πρότυπα. Πρέπει να πετήσουμε τα πιο υψηλά πρότυπα του ελέγχου της μετανάστευσης και της δημόσιας ασφάλειας. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να διευκολύνουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο για την εισρωή νόμιμων ροών στην επικράτειά μας. Ο στόχος αυτός είναι βασικό στόχος και το συμμεριζόμαστε πλήρως και η διευκόλυνση των διαδικασιών και η ελάφρυνσή του, η ελάφρυνση του άκτους μας οδηγεί στο να ζητήσουμε ότι το άτομο να μην την ώρα που ζητά την ε, έκδοση της θεώρησης να είναι παρόν Φυσικά να έχουμε φυσική παρουσία, επίση να αυξήσουμε το κριτήριο τη νομική ασφάλεια, τη ασφάλεια δικαίου, τη μείωση των προθεσμιών και τη δυνατότητα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία για την έκδοση των θεωρήσεων. Τώρα, ένα άλλο σχόλιο σε σχέση με το θέμα τη ασφάλεια, και εδώ πρέπει να είμαι πολύ σαφή. Η διευκόλυνση έκδοση θεωρήσεων δεν έχει να κάνει με τη χαλάρωση των κριτηρίων περί ασφάλειας. Όπως ε, είδαμε στην ε, εξέταση της διαδικασίας, ε, πολλές φορές έχουμε το τυχαίο και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ταχεία και αποτελεσματική έκδοση θεωρήσεων. Δεν υπάρχει τίποτα στην πρόταση που να μπορεί να θεωρηθεί ότι υποσκάπτει την ασφάλεια. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων, για την υποβολή της αίτησης και της απόκτησης της θεώρησης. Αυτό είναι σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Λεγθέντως αυτού, θα σχολιάσω ορισμένες τροπολογίες που εγώ έχω εισαγάγει και έχω συμπεριλάβει και τις προτάσεις πολλών συναδέλφων για να αποσαφενήσω την πρόταση αυτή της Επιτροπής για το ποια μορφή πρέπει να πάρει ο κώδικας θεωρήσεων. Καταρχήν, οι τροπολογίες ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας, δηλαδή να έχουμε μια ορθολογική διαδικασία, να έχουμε ένα ηλεκτρονικό φάκελο όπου να περιλαμβάνονται η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και να μην χρειάζεται με το χέρι να συμπληρώνονται τα έγγραφα. Έτσι λοιπόν τα προξενία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικά να δέχονται αιτήσει. Τώρα, το σημείο 6.1α για τις προθεσμίες. Ήθελα να ενισχύσω τους στόχους ε, της πρότασης περνώντας από τους 6 στους 9 μήνες για την προθεσμία. Γιατί τώρα εδώ αλλάζει τον μοντέλο των ταξιδιών, δηλαδή όλο ένα και περισσότερο χρόνο πριν κανονίζει κάποιος ε, το ταξίδι του και αγοράζει τα εισιτήρια. Έτσι λοιπόν, ε, νομίζω ότι είναι λογικό να έχουμε νέα αντί για έξι μήνες στην προθεσμία. Επίσης υποστηρίζω το να δίνονται οι περισσότερες θεωρήσεις ε, πολλαπλών εισόδων. Νομίζω ότι αυτό ε, διευκολύνει και τα προξενία αλλά και τους ετούντες και ε, πρέπει να εξυγχρονίσουμε το VIS, το σύστημα θεωρήσεων. Πρέπει να διευκολύνουμε τους ταξιδιώτες που είναι καλοί τυπίστη και πρέπει να καταστήσουμε πιο ευέλικτο τον ορισμό αυτής της κατηγορίας ταξιδιωτών. Παραδείγματο χάρη, ε, μέσα στους 18 μήνες να έχουν χρησιμοποιήσει δύο φορές τη θεώρηση άνθρωποι αυτοί, αντί για 12 μήνες όπως έχουμε στην πρόταση της Κομισιόν. Και πολύ συνοπτικά θέλω να φέρω ένα θέμα υψηλής ευαισθησίας. Πρόκειται για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις όπως αποκαλούνται. Ξεκινάμε από τη βάση ότι αυτή η φόρμουλα ε, δεν λύνει την τεράστια πρόκληση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει με τους ετούντες άσυλο. Και επίσης, καθώς ε, αυτή είναι μια συμπληρωματική οδός παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι μειοδός που θα πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη όταν θα διευκολύνουμε την σίγουρη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρώπων που ε, ουσιαστικά διώκονται και θέλουν να αποφύγουν τον πόλεμο. Εδώ μιλάμε για κάτι που είναι απαραίτητο να το προωθήσει αυτή η Επιτροπή, καθώς βλέπουμε μια τεράστια έξοδο και φυσικά υπάρχει και αναγκαιότητα να συμπληρωθεί η ανθρωπιστική θεώρηση και με άλλα μέσα. Τώρα εδώ πρέπει να δράσουμε ως συνομοθέτες μαζί με το Συμβούλιο. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να το κάνουμε, αν όχι τώρα πότε. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι νομοθέτες έχουμε την υποχρέωση να ανοίξουμε το παράθυρο σε μια δυνατότητα ανθρωπιστικής θεώρησης που να διευκολύνει την έκδοση της θεώρησης και την δυνατότητα νόμιμης πρόσβασης στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι άνθρωποι έρχονται από τόσο ταλανισμένες περιοχές όπως βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα. Και την περασμένη Πέμπτη, με αυτό το πνεύμα υιοθέτησε το Κοινοβούλιο το ψήφισμά του για την κρίση των προσφύγων. Ουσιαστικά ε, μιλούσε εκεί για την εισαγωγή ανθρωπιστικών θεωρήσεων μέσω της τροποποίησης του κώδικα θεωρήσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή η Επιτροπή να κάνει τα περιτευμένα για να βρει τα κατάλληλα τον κατάλληλο τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα. Τώρα θέλω να προσθέσω και την προβληματική που έχει να κάνει με την μεταχείριση των συγγενών ε, των πολιτών από τρίτες χώρες. Πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να επισκεφτούν τους συγγενείς τους και γι' αυτό ζητούν θεώρηση. Μιλάμε για παππούδες που θέλουν να επισκεφτούν τα εγγόνια τους ε, ή παραδείγματος χάρη για παιδιά χωρισμένων γονιών που θέλουν να επισκεφτούν τους γονείς τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή του κώδικα θεωρήσεων ε, πολλές φορές ε, καταλήγει σε κάποιες απορρίψεις που δεν θεμελιώνονται όπως πρέπει και η οδηγία 2004-38 δίνει δικαίωμα σε θεώρηση σε ε, κατοίκους τρίτων χωρών που ε, έχουν συγγενείς που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως σε περιπτώσεις αρνήσεων ποτέ δεν αιτιολογούνται επαρκώς. Φαίνεται ουσιαστικά αυτές ε, οι απορρίψεις να αιτιολογούνται βάση του εγχειριδίου και όχι βάση του ίδιου του κώδικα θεωρήσεων. Δηλαδή ουσιαστικά η εφαρμογή των κανόνων γίνεται τυχαία και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν για να ενισχύσουμε ορισμένες διατάξεις. Πέρα από το θέμα της διαδικασίας που έχει να κάνει με ε, το να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στα προξενία χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει τέλη, θα πρέπει και να υπάρχει λεπτομερής αιτιολόγηση όταν απορρίπτεται το αίτημα της έκδοσης θεώρησης από τα προξενία για να γνωρίζουν τα άτομα γιατί έχει υπάρξει η άρνηση αυτή της έκδοσης θεώρησης. Άρθρο 18. Και επίσης ε, θα πρέπει εδώ να δούμε και το θέμα των προσφυγών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια καλή εικόνα προς το εξωτερικό για να ενισχύσει και την έκδοση θεωρήσεων Σένκεν. Θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε και μία ιστοσελίδα ε, που τουλάχιστον ε, να υπάρχει σε πέντε επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών, άρθρο 45. Επίσης τώρα θέλω να αναφερθώ και στους εργολάβους, στους ε, εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, το θέμα της εξωτερικής ανάθεσης της υπηρεσίας. Σίγουρα ο όγκος ε, των αιτήσεων μας οδηγεί στο να χρησιμοποιούνται συχνά αυτές ε, οι επιχειρήσεις. Όμως εδώ μιλάμε για πληροφορίες ευαίσθητου περιεχομένου και γι' αυτό χρειάζεται να τροποποιηθεί το άρθρο 38 που έχει να κάνει με το θέμα του outsourcing, την εξωτερικής ανάθεσης. Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση από την πλευρά της Κομισιόν και να εφαρμοστούν όλες οι εγγύσεις για αυτούς τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Επίσης, το θέμα της ε, υποχρεωτικής εκπροσώπησης από ένα τρίτο κράτος όταν δεν υπάρχει προξενική εκπροσώπηση σε ένα κράτος μέλος προτείνω ένα νέο άρθρο για κέντρα θεωρήσεων Σέγγεν και να ενισχύσουμε την προξενική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για να διασφαλίσουμε το στόχο αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα εδώ να μπούμε σε διοργανικές διενέξεις σε σχέση με το πώς θα αναπτυχθεί ο σημερινό κώδικα θεωρήσεων, αλλά θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ με την προσέγγιση τη Κομισιόν μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων μετέπειτα να παραπέμψει ε, και να υλοποιήσει την κατάρτιση των παραρτημάτων. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δουν οι συνομοθέτες, όχι να έχουμε εδώ κατεξουσιοδότηση πράξης. Αυτά προς στιγμή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τον συμπληρωματικό χαρακτήρα αυτού του φακέλου σε σχέση με την θεώρηση περιοδίας. Ο κύριος Σορτφέ είναι ο αρμόδιος εισηγητής για το θέμα αυτό και φυσικά θα πρέπει η έκθεση αυτή να φέρει ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα με τη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ. Thank you. Now uh, uh, uh, Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε χρόνο τώρα για τους και Και σπέκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω ευθύ εξ αρχή ότι είναι πολύ ωραίο και ευχάριστο ότι, ο συνάδελφος Λόπε Αγγιλάρη είναι μαζί μας και μαχητικός στο ring έτοιμος. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επίσης μας παρουσίασε κάποιες σημαντικές πτυχές αυτού του θέματος. Σας ευχαριστούμε για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, σας ευχαριστούμε επίσης γιατί τίθενται οι στόχοι του τουρισμού της ενδυμάμωσης ε, του τουρισμού στην Ευρώπη, κάτι που πραγματικά μπορεί να μας δώσει πολλές θέσεις απασχόλησης και πολλές ευκαιρίες. Ε, ενδυνάμωση της απασχόλησης εντός και εκτός της Ευρώπης. Αυτή η στόχη είναι για μας πολύ σημαντική. Θεωρώ λοιπόν σημαντική την πρωτοβουλία. Και να σας αναφέρω και κάποια σημεία. Πολύ θετικό είναι αυτό που ο συνάδελφος μόλις παρουσίασε, δηλαδή η περισσότερη ευελιξία των εξωτερικών φορέων παροχής υπηρεσιών. Εδώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της απόστασης των 500 χιλιόμετρων από τον τόπο διαμονής κτλ. λοιπά, Δηλαδή το θέμα επίσης των προξενικών αρχών και των αρμοδιοτήτων και ευθύνης τους. Εγώ βεβαίως ε, έχω κάποιες ε, συγκεκριμένες προτάσεις για τροπολογίες. Το θέμα ε, της πρότασης για τις βίζες Σέγγεν δεν είναι κάτι που να το δω πολύ θετικά. Επίσης το θέμα της ασφάλειας και του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς καμία δικαιολογία απέρριψε την ε, ασφάλεια για θέματα ασθένειας. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει ίσως να ξανασκεφτούμε, να επεξεργαστούμε κάποια άλλα σημεία, όπως παραδείγματο χάρη την υποχρέωση οι προξενικές αρχές immediately όπως λέει το κείμενο, άμεσα δηλαδή ε, να θέτουν προθεσμίες. Αυτό μου φαίνεται λίγο άκαμπτο και νομίζω δεν πρέπει εδώ να περιορίσουμε υπερβολικά τις δυνατότητες των ε, προξενείων. Ίσως να πούμε ε, θα έπρεπε, θα μπορούσαν, δηλαδή η διατύπωση δεν μπορεί να είναι τόσο περιοριστική. Αυτή θα είναι μια άλλη τροπολογία που ίσως υποβάλλω. Το θέμα των 15 ημερών 15 ημέρες για ένα μόνο κράτος. Μα κοιτάξτε, βεβαίως πρέπει να υπάρχει ε, πάντα το θέμα της ασφάλειας το οποίο θα διέπει τις ε, προτάσεις. Αλλά, αλλά αυτό το 15 ημέρες για μια χώρα μου φαίνεται ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε. Το θέμα τώρα της ανθρωπιστικής βίζας όπως τη λέμε, ανθρωπιστικής θεώρησης. Η θέση του ΕΛΚ είναι εδώ ότι αυτή η ανθρωπιστική βίζα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει για να είναι κατανοητή εδώ η πρόταση αυτή θα πρέπει να την επεξεργαστούμε περαιτέρω και εδώ χρειάζονται σαφώς κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποίησεις στο δίκαιο που αφορά το άσυλο. Είναι κάτι που οπωσδήποτε έχει σχέση με το θέμα του ασύλου. Αυτοί δηλαδή που ζητούν άσυλο και βεβαίως και τα προγράμματα μετεγκατάστασης και όλα τα, όλες οι συναφείς διατάξεις. Καταλαβαίνω ότι εδώ βεβαίως εξαιτίας των ε, πρόσφατων γεγονότων και της επικαιρότητα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Αυτή η έκθεση σίγουρα θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και σίγουρα θα προετοιμάσω και εγώ τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ ε, όλους για την εργασία τους. Ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ στον, τον εισηγητή για την θετική αξιολόγηση της πρότασης της Κομισιόν. Όπως λέμε και στο επεξημενικό σημείωμα, ε, διευκολύνουμε τους νομιμούς ταξιδιώτες και απλουστεύουμε και το νομικό πλαίσιο για τα πραξενία των κρατών μελών. Αυτά τα τόνισε και ο εισηγητής καθώς και το θέμα της προστασίας από την παράτυπη μετανάστευση. Υπάρχει όμως και ένας άλλος επιπλέον στόχος για την Κομισιόν. Είναι το θέμα της οικονομικής πρόοδου. Ως προς τα συγκεκριμένα σχόλια τώρα για τις τροπολογίες. Πρώτον, όσον αφορά την δυνατότητα ηλεκτρονικών διαδικτυακών αιτήσεων. Είμαστε υπέρ, γιατί εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε την υποβολή των αιτήσεων, όμως να διακρίνουμε την συμπλήρωση της αίτηση επιγραμμικά, διεκτυακά, από την υποβολή από οπουδήποτε, το οποίο δεν γίνεται για τεχνικούς λόγους. Είναι θέμα συμπλήρωση του εντύπου το οποίο πρέπει να επιστραφεί αυτό καθ' αυτό. Σε μερικέ χώρες μάλιστα το διαδίκτυο δεν λειτουργεί τόσο οικονομικά και πρέπει να προσφύγουμε, να καταφύγουμε τελικά στο χαρτί και την υπογραφή. Ε, και λοιπόν στο σύστημα αυτό θα καταγράφονται οι ταξιδιώτες, αυτό μας βρίσκει σύμφωνο, το είπε και ο βεβαίω. και θέλω να διακρίνουμε του καλή πίστη ετούντες που είναι τακτικοί ταξιδιώτες από αυτούς που ταξιδεύουν για πρώτη φορά. Διαφορετικό. Γιατί εδώ μιλάμε για θεώρηση πολλαπλών εισόδων. Ε, το θέμα που μας αφορά εδώ πέρα είναι αυτοί που υποβάλλουν έτσι για πρώτη φορά. Πάντως είμαστε υπέρ αυτής της προσέγγισης. Θέλουμε να ορίσουμε αυτές τις κατηγορίες με πιο ευέλικτο τρόπο ε, και να επεκτείνουμε την περίοδο των 12 μηνών σε 18. Αυτό πιστεύω ότι είναι εύκολο να ρυθμιστεί. Θα καταλήξουμε σε μια συμβαστική συμφωνία. Όσον αφορά την θεώρηση για ανθρωπιστικού λόγου, οι τροπολογίε, οι σχετικέ τροπολογίε ε, ε, έχουν κάποια κριτήρια, α πούμε τη διεθνή προστασία. Να υπάρχει λοιπόν και εδώ η δυνατότητα έκδοση θεωρήσεων με περιορισμένη γεωγραφική ισχύ, ακριβώ για να μπορέσουμε να παράσχουμε την διεθνή προστασία σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η Κομισιόν ήδη έχει εκφανθεί από αυτού. Είναι υπέρ του στόχου. Κατανοούμε ε, ασφαλώ γιατί ο εισηγητή προτείνει ότι προτείνει, ιδιαίτερα εν ώψη τη τραγική κατάσταση στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, ο κώδικα θεωρήσεων ενδεχομένω δεν είναι το καταλληλό εργαλείο για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Ακούστηκαν και άλλες προτάσεις. Ε, το θέμα της ε, μετεγκατάστασης, για παράδειγμα, θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Αρκεί να γίνει εγκαίρος βεβαίως για να προστατεύσουμε αυτούς που πρέπει να προστατεύσουμε. Και έχουμε και το πακετό θεωρήσεων, το Visa Package, το οποίο και αυτό πρέπει να το δούμε κατεπηγόντως. Από την άποψη αυτή, η Κομισιόν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την ε, μετανάστευση έχει υποβάλει πολλές προτάσεις είναι την περισμένη εβδομάδα ε, όσον αφορά την μετακατάσταση η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτός είναι πλέον κατάλληλο κατάλληλος τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα. Για καταρχήν 20.000 πρόσφυγες. Το πόσο αυτό έχει ο, το αριθμός αυτός έχει ήδη αυξηθεί, η Κομισιόν υπέρ αύξηση του πλήθους αυτού. Ο μηχανισμός αυτός προβλέπει εθνικές αποφάσεις έγκρισης εισδοχής. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία σε σχέση με την θεώρηση περιορισμένης γεωγραφικής ισχύω που αναφέρατε στην τοπολογία. Όσον αφορά τη συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, η Κομισιόν συμφωνεί με τον εισηγητή ότι η εκχώρηση αυτών των καθηκόντων εκεί που δεν υπάρχουν και τα προξενία θα βοηθήσει τους α, ε, ταξιδιώτες. Και μπορούμε έτσι να κρατήσουμε τα έξοδα χαμηλά, αν και κάποιος ενδεχομένω να χρειαστεί να ταξιδέψει από πόλη σε πόλη. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία με τρίτους, με εξωτερικούς εργολόγους, ε, οι οποίοι όμως δεν έχουν ευθύνη επιλογής ή έγκρισης, μόνο θα συλλέγουν τα στοιχεία και θα τα μεταφέρουν, θα μεταδίδουν στην Κομισιόν. Ενώ ότι δεν εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης της ε, θεώρησης, αυτό παρακαλώ να το σημειώσετε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σημειώστε επίση ότι η εφαρμογή των άρθρων που αφορούν τους εξωτερικούς εργολάβους περιέχει επίση ε, ρήτρα περί συνεχούς αξιολόγησης. Θα χρειαστεί λοιπόν να επιβάλλουμε κάποια τροπολογία εκεί στο ή στα σχετικά άρθρα. Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, η Κομισιόν χαίρεται για την υποστήριξη της ιδέας της πολιτική εκπροσώπησης, παρουσίας μάλλον, και όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης των κέντρων υποβολής αιτήσεων, θα συνεργαστούμε με τα κρατημέλη βάσει τη αξιολόγηση και των διατάξεων του παροντό κώδικα θεωρήσεων. Είμαστε ω Κομισιόν υπέρ μια πιο ευέλικτη προσέγγιση του θέματο. Πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Θα χρειαστεί, όμω ένα πλαίσιο συνεργασία με τα κράτη-μέλη και θα δούμε ποιο είναι και ο καταλληλότερο μηχανισμό συνεργασία, λαμβάνοντα υπόψη των κρατόπου συνθήκων. Όπω είπα, προτείνουμε για όλους αυτούς τους λόγους μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Ε, Δυστυχώ οι προτάσει του ΣΥΤΗ δεν έχουν πετύχει το απαιτούμενο, το επιθυμητό αποτέλεσμα, γι' αυτό και θα γίνουν κάποιε τροποποιήσει στην πρόταση. Τέλο, και εν συντομία, όσον αφορά τι τροπολογίε που αφορούν την διαγραφή των ε, επιχειρησιακών παραρτημάτων και την έγκριση των εφαρμοστικών αποφάσεων, εμεί θα προτιμούσαμε να τα διατηρήσουμε τροποποιώντα τι κατεξουδότερε πράξης. Το εξετάσαμε πολύ προσεκτικά να ξέρετε, είδαμε το γενικότερο πλαίσιο και όχι, είναι επιχειρησιακά απαιτητά αφορούν την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ε, σχετικά με το πώ δηλαδή συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι καθαρά επιχειρησιακά θέματα. Λοιπόν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε, τα χρειαζόμαστε. Το ίδιο για την θεώρηση που Χάμπουργκ. Αυτά θα τα ρυθμίσουμε στις εφαρμοστικές αποφάσεις. Αυτά ως πρώτα σχόλια στις τροπολογίες, στις προτάσεις τροπολογίες του ECT. Ευχαριστώ τον ίδιο και τον Σκιώδη για τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθυνθώ στην Προεδρία του Λουξεμβούργου για να αντιδράσει. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Εξαιρετικά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ που μείνετε το λόγο. Η, πρόεδρα, η Προεδρία διάβασε την ε, πρόταση τη Επιτροπή και θυμίζω βεβαίω και την έκθεση του εισηγητή του κ. Λόπε Αγγιάρη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ οικονομική ανάπτυξη, ελευθερία κίνηση και προστασία των ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν μια συζήτηση προσανατολισμού στο Συμβούλιο ΖΑΙ του Οκτωβρίου έτσι ώστε να επιταχύνουμε τις εργασίες στην ομάδα εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής θέλει να κάνει μια σύντομη σύνοψη. Σύντομη. Όχι, ναι. Πολύ σύντομα. Εγώ άκουσα την επικοδομητική θέση που εξέφρασε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ και φυσικά αφού άκουσα και το Συμβούλιο και την Κομισιόν πρέπει απλώς να υπογραμμίσω το εξή. Η πρόθεση του εισηγητή είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για την έκδοση των θεωρήσεων, ε, φυσικά διαφυλάσσοντας τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια δικαίου. Γι' αυτό ακριβώ επιμένουμε στην αναγκαιότητα να αιτιολογούνται όπως πρέπει οι απορρίψεις, κυρίως ε, ό,τι έχει να κάνει με τις θεωρήσεις που ζητούνται από συγγενείς. Γιατί ουσιαστικά αυτό λέγεται στον κώδικα θεωρήσεων. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία και ελπίζω να τη βρούμε στη συζήτηση στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 25 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα θα περάσουμε στη θεώρηση περιοδίας. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν στον εισηγητή, τον κύριο Ορτφέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Introduit de par rapport à la position de la. Ευχαριστώ. Θα σας ε, παρουσιάσω το θέμα αυτό μετά από τις ανταλλαγές απόψεων που είχαμε την Άνοιξη με την Επιτροπή αλλά και μετά <clears throat> την επίσκεψη που κάναμε στην Κωνσταντινούπολη με μέλη της Επιτροπής. Πρόκειται για το θέμα της θεώρησης περίγησης, ένα καινοτόμο εργαλείο, ένας τρόπος να δημιουργηθούν από 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις ευρώ το χρόνο. Ε, αυτό είναι στοιχεία που μας έχει δώσει η Επιτροπή, χωρίς βεβαίως να έχουμε απολύτως καμία απόδειξη αυτή, αυτή τη στιγμή. Ε, πρόκειται για κάτι το καινοτόμο, καθότι από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει απολύτως καμία τέτοια περίπτωση θεώρησης, βίζας που να επιτρέπει σε κάποιον να περιηγηθεί σε περίπου 10 χώρες επί πολλούς μήνες και βεβαίως ε, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η ε, νέα διαδικασία, ποιες είναι οι αδυναμίες και γι' αυτό και προτείνω να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα σας εξηγήσω γιατί. Οι τουριστικές περιηγήσεις στην Ευρώπη είναι συχνά ενδοευρωπαϊκές. Το 83-84% παραδείγματος χάρη των τουριστών στην Γαλλία ήταν Ευρωπαίοι. Οι υπόλοιποι ήταν σε μεγάλο βαθμό Αμερικανοί, Ασιάτες και αυτό ισχύει και για τις περισσότερες χώρες. Βλέπουμε ότι 582 εκατομμύρια τουρίστες είναι το τελευταίο νούμερο για το 2014 και διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται κατά 15 εκατομμύρια παραδείγματο χάρη τον τελευταίο χρόνο και μάλιστα η προβλέψη είναι να φτάσει τα 744 εκατομμύρια τουρίστες. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη που σήμερα εκδίδουν αυτές τις ε, θεωρήσεις, όπως παραδείγματο χάνει διάφορες ε, αρχές ε, στην Ευρώπη, στη Γαλλία παραδείγματος χάρη, το κάνουν για να διευκολύνουν αυτές τις τουριστικές επισκέψεις. Σήμερα μιλάμε λοιπόν για μια ευρωπαϊκή θεώρηση η οποία θα επιτρέπει ελεύθερη κυκλοφορία σε όλο το χώρο Σέγγεν χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου ή παρακολούθησης αυτών ε, των μετακινήσεων. Ένας τουρίστας σήμερα βεβαίως μπορεί να ε, δικαιολογήσει αυτές τις μετακινήσεις τους και ξέρουν σήμερα πολύ καλά οι προξενικές αρχές πόσο επιφυλάσσονται, ξέρουμε σήμερα πόσο επιφυλάσσονται, να εκδώσουν τέτοιου είδους ε, θεωρήσεις περιήγησης, καθότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Για κάποιες βεβαίως κατηγορίες, όπως οι αθλητές, είτε οι καλλιτέχνες, αντιμετωπίζουν σήμερα πολλά εμπόδια, διοικητικά και άλλα. Η βίζα λοιπόν περιήγησης δικαιολογείται εάν είναι πλαισιωμένο και δεν υπάρχουν καταχρήσεις ε, για διάφορους λόγους. Θα σας παρουσιάσω εδώ τα σημεία αυτά της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απαιτούν κάποιες εγγύησεις έτσι ώστε ο ετών να μπορεί να οργανώσει τις ε, περίγεις του. Και θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής που θεωρεί ότι η χώρα στην οποία μπαίνει καταρχήν ο ετών θεώρηση θα πρέπει να την εκδώσει και για τις υπόλοιπες χώρες. Το θέμα λοιπόν είναι εδώ εάν θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ της χώρας Α και της χώρας Β. Μου φαίνεται ότι η αρμόδια χώρα για την εξέταση είναι η χώρα αυτή στην οποία θα διαμείνει και θα ασκήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο ετών και όχι η χώρα εισόδου. Θα πρέπει να δίνεται μία ε, λίστα, ένας κατάλογος που να καλύπτει όλες τις κατηγορίες. Εγώ προτείνω ο κατάλογος αυτός να περιλαμβάνει τις κατηγορίες τις επαγγελματικές. Σε ποιους δηλαδή επαγγελματίες θα ε, δίδεται μία τέτοια βίζα περιήγησης. Όσον αφορά την διάρκεια, 181 ημέρες, και βεβαίως θα πρέπει να υποβάλλονται και πιστοποιητικά για την διαδρομή, για τον λόγο, τον επαγγελματικό της περιήγησης, για καλλιτέχνες, για αθλητές, καθώς και για τους οργανισμούς οι οποίοι οργανώνουν αυτήν την περιήγηση ή προσκαλούν τον καλλιτέχνη ή τον αθλητή. Ο υπεύθυνο οργανισμός θα πρέπει λοιπόν εδώ να εγγυάται με ένα πιστοποιητικό την αίτηση. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται και η σύμβαση εργασίας, η ύπαρξη και τα δικαιολογητικά για μια ασφάλεια η οποία να αναγνωρίζεται και να ισχύει σε όλες τις χώρες στις οποίες θα διαμείνει ο ετών, άδεια διαμονής, άδειες εργασίας για όλες τις χώρες στις οποίες θα εργαστεί ο ετών και βεβαίως η ελευθερία κίνηση στο εσωτερικό του χώρου Σέγγεν απαιτεί αυτές τις εγγύσεις για μια θεώρηση, για μια συγκεκριμένη διαμονή. Καταλαβαίνετε ότι σε κάθε περίπτωση Πρόκειται για μία κυκλοφορία που ξεπερνά τους τρεις μήνες και αφορά πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποία ο ετών θα μπορέσει να ασκήσει μια επαγγελματική δραστηριότητα. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει και μία χρονική περίοδος των 30 ημερών, καθότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ε, διενεργήσουν ελέγχους. Οι αιτήσει θα πρέπει να υποβάλλονται 6 μήνες πριν την άφηξη και 3 μήνες ή 2 μήνες το αργότερο πριν από την άφηξη. Αυτό δικαιολογείται από την διάρκεια προετοιμασίας και είναι πολύ σημαντικό να μην λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, κάτι που θα οδηγούσε σε περισσότερες αρνητικές απαντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να μπορούν να ελεγχθούν οι οργανισμοί που δικαιολογούν και επιστοποιούν την αίτηση, την αξιοπιστία τους και καταλαβαίνετε ότι οι προξενικές αρχές δεν μπορούν να διενεργήσουν όλους αυτούς τους ελέγχους μέσα σε 20 ημέρες. Είναι λοιπόν αδύνατον να τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, γι' αυτό και ζητούμε μεγαλύτερη διάρκεια, καθότι αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρξει έλεγχος σε περισσότερες της μίας χώρες. Τώρα, για επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στις χώρες Σέγγεν, επί ένα χρόνο βλέπετε ότι εδώ προτείνουμε το αντίτιμο των 60 ευρώ. 60 ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 90 δολάρια. ...136 δολάρια πάντα στις, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς προτείνουμε λοιπόν εδώ ε, 100, όσο είναι δηλαδή και το αντίτιμο για ένα διαβατήριο ευρωπαϊκό, καθώς και 50 ευρώ επιπλέον για την ε, επιμήκυνση της ε, διάρκειας ισχύω αυτού του εγγράφου. Ακόμα δεν υπάρχουν βεβαίω παρά μόνο διμερείς ε, συμφωνίες. Κανείς όμως δεν ξέρει ποιες είναι οι χώρες που θα προσχωρήσουν από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε από μέρους των τρίτων χωρών. Δεν γνωρίζουμε τις συμφωνίες, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη να αντιτεθεί σε συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια κάτι που μου φαίνεται επικίνδυνο. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για χώρες Σέγγεν όπως η Ελβετία, δηλαδή συμπεριλαμβάνονται η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία σε αυτές. Αν λοιπόν καταργηθούν αυτές οι ιστορικές συμφωνίες, θα υπάρξουν ενδεχομένες και αντίπεινα από μέρους αυτών των τρίτων χωρών. Αυτή λοιπόν η βίζα περιήγησης και για πολλούς άλλους λόγους θα μπορούσε να είναι αντικείμενο συζήτησης. Νομίζω ότι σας έχω εκθέσει εδώ τους πιο σημαντικούς, αλλά βεβαίως θα πρέπει η ε, συζήτηση να συνεχιστεί. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και θα σημειώσω όλα σας τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Λόπες Αγγιλάρ. Ο ευχαριστώ, Πρόεδρε Εκνέου και ευχαριστώ και τον κύριο Ορτφέ για την παρουσίαση της έκθεσης ε, για αυτή την ε, λεγόμενη Touring Visa την ε, θεώρηση περιήγησης και εγώ είμαι σκιώδης για τους σοσιαλιστές όπως ξέρετε και, στον κωδικα, και ο κωδικας θεωρήσεων και αυτή η θεώρηση αποτελούν ένα πακέτο. Το υπογράμμισα προηγμένως ε, γιατί θέλουμε να εγγυθούμε την ε, συνοχή της γενικής προσέγγισης στην ε, δημιουργία της κοινοτικής πολιτικής μέσω αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας που φύγει και τα δύο αυτά στοιχεία του πακέτου. Υπάρχουν ε, πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Σορτφέ που μου φαίνονται θετικά, όμως θα αναφερθώ σε αυτά τα σημεία που προκαλούν ανησυχία στην ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών. Αυτό γιατί αναφέρονται στην ε, θέση που εξέφρασε ο εισηγητής, ε, δηλαδή ε, να έχουμε ένα, διευρυμέ, ένα πιο στενό πεδίο εφαρμογής για να περιλάβουμε εκεί τους καλλιτέχνες και τους αθλητές. Αναφέρομαι στην τροπολογία 15 αφήνοντας εκτός άλλες κατηγορίες που θα μπορούσαν να ωφεληθούν και που αναφέρονταν στην πρόταση της Κομισιόν και συμπεριλαμβάνονταν φυσικά όχι μόνο οι αθλητές και οι καλλιτέχνες αλλά και οι συνταξιούχοι τουρίστες που κάνουν ε, κάποιες ε, επισκέψεις διαρκείας ή ε, παραδείγματος χάρη τους αλλοδαπούς φοιτητές οι οποίοι παραδείγματος χάρη ταξιδεύουν για να κάνουν ένα μάστερ και στη συνέχεια επισκέπτονται και άλλες χώρες πέρα από τη χώρα στην οποία υλοποίησαν τις σπουδέ τους. Και φυσικά και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, η πρόταση του κυρίου Ορτφέρα αλλάζει την αρχική πρόταση της Κομισιόν γιατί επιβάλλει περισσότερες προϋποθέσεις στους ετούντες, τροπολογία 36. Εδώ έχουμε το εξή παράδοξο ενώ θέλουμε να διευκολύνουμε την έκδοση θεωρήσεων, προκειμένου να ευνοήσουμε τους ταξιδιώτες καλή την πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν η ιδέα, βρίσκουμε εδώ τελικά ένα πρόσθετο εμπόδιο ή μια δυσκολία, αν θέλετε, και εμείς δεν συμφωνούμε ως σοσιαλιστές με τη φιλοσοφία αυτή. Επίσης διαπιστώνω ότι μειώνεται ο χρόνος διάρκειας της ε, θεώρησης αυτής, καλωθώς και η ε, δυνατότητα να παραταθεί ένα χρόνο σε 60 ημέρες. Αυτό στην τροπολογία 63. Και τέλος παρατηρώ ότι δημιουργείται μια διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών που θα ε, αποφασίσουν ότι η νέα θεώρηση δεν θα πρέπει να καθιστά άκυρες τις εθνικές θεωρήσεις. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε όμως για ένα συμπληρωματικό εργαλείο. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε μια θεώρηση στις εφιστάμενες εθνικές θεωρήσεις. Είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας για να μελετήσουμε την έκθεση εις βάθος, όμως ε, θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί απέναντι σε αυτό το όρομα που παρουσίασε ο κύριος Ορτφέ και ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, να βρούμε κάποιες λύσεις για να οδεύσουμε προς την αρχική πρόταση της Κομισιόν και να πετύχουμε μια χρήσιμη συμφωνία επί της έκθεσης αυτής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Τομάσικ. Ευχαριστώ. Το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκει σύμφωνος ως ομάδα διότι προσελκύουμε έτσι ξένες επενδύσεις και τουρισμό υπέρ των ευρωπαϊκών οικονομιών. Εν τούτης, υπάρχουν κάποια επιμαχά σημεία. Πιστεύουμε συγκεκριμένα ότι το μέτρο θα προσελκύσει περισσότερο τουρισμό και επενδύσεις όπως προείπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελέτες δείχνουν συνεχώς ότι η δυσκολία να τα βγάλει κανείς πέρα με το σημερινό σύστημα αποτρέπει επισκέπτες από τον έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά υπάρχουν και τα θέματα ασφάλειας. Πρέπει λοιπόν το σύστημα να συνάδει, να συντονίζεται, να συνεργάζεται με τα συστήματα ασφαλείας και με το SIC και το VIC, το σύστημα επεξεργασίας θεωρήσεων. Και υπάρχει ένα σαφές σύστημα δυνατοτήτων, τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν εξαιρέσει, απαλλαγές να μην διορθώνω και να μην ε, υπάρχει δυνατότητα το κάθε κράτο να κάνει ό,τι θέλει με εξαιρέσει. Οι ίδιοι κανόνε δεν ισχύουν έναντι όλων με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δεπρέ. Παρακαλώ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, άργησα στην Επιτροπή Προπολογισμών. Είχαμε και μια έκθεση όσον αφορά τα κονδύλια τα οποία θα δοθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του χρόνου. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά συζητήσαμε ως τώρα, παρουσιάσαμε τουλάχιστον τις δύο εκθέσεις του κ. Τεφέ, κυρίως, και ξεκινώ από τις θεωρήσεις περιήγηση. Εξαιρετική δουλειά, πρώτα απ' όλα, επί συγκεκριμένων σημείων να σας πω τις απόψεις μου. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή καταρχάς. Θεωρώ ότι όσον αφορά ένα νέο σύστημα, ένα νέο μηχανισμό δεν έχει ισοδυναμό γιατί ως τώρα ο τύπος αυτός θεώρησης δεν υπήρχε. Όσον αφορά λοιπόν το πεδίο εφαρμογή, το αντικείμενο, καλό θα ήταν να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί παρά εκτατικοί, στην αρχή τουλάχιστον. Γιατί θα χρειαστεί μια αξιολόγηση κάποια στιγμή γιατί μπορεί να διαπιστώσουμε ότι είναι αντικείμενο κατάχρηση κλπ. Είναι δύσκολο να κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω. Είναι πολύ πιο εύκολο να διευρύνουμε το αντικείμενο παρά να κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω από τη στιγμή που έχουμε συμπεριλάβει μια κατηγορία δικαιούχων. Θα έλεγα λοιπόν, α είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι στην αρχή, αν θέλετε, όσον αφορά τι κατηγορίε των πιθανών δικαιούχων. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε Ποιε εγγυήσει μπορούν να μα παράσχουν όσον αφορά την παραμονή στο σημείο Α, στη χώρα Β κλπ. Τώρα για του καλλιτέχνε, του αθλητέ. είναι σαφέ. Ε, ε, για του τουρίστε τα πράγματα είναι πολύ πιο ασαφή. Δεν είναι ότι πηγαίνει ο ε, σε ένα στάδιο συγκεκριμένο ή ο ηθοποιό σε ένα θέατρο. Ε, δεν θέλω να μα περιορίσω για το μέλλον, αλλά για την αρχή τουλάχιστον παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι όπω είπα να μην ξενυχτούμε πολύ από την αρχή. Καλό θα είναι λοιπόν να περιοριστούμε στην αρχή πρώτα. της Κομισιόν. Ναι λοιπόν για τους αθλητές, ναι για τους καλλιτέχνες. Να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για τα στελέχη επιχειρήσεων κλπ. Σύμφωνοι μέχρι εκεί ναι. Για τους, και για τους φοιτητές ενδεχομένως, στα πλαίσια πανεπιστημιακών ανταλλαγών. Εκεί υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, ε, δεν χρειάζεται ο συγκεκριμένο διάβλο. Τώρα, όσον αφορά τις προϋποθέσεις παράτασης. Η ιδέα του κ. Ερτοφέ είναι καλή. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή, να το συζητήσουμε. Όμως, η ιδέα, η πρόταση, η διάρκεια της θεώρησης, να μπορεί να παραταθεί λίγο περισσότερο από τη διάρκεια της απασχόλησης, πούμε, για κάποιους μήνες ενδεχομένω, σύμφωνοι. Το κριτήριο που προτείνει ο ασχητής είναι σωστό. Τώρα όσον αφορά την παράταση της διάρκειας, προβλέπετε εδώ τι. Μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο, την προκαθορισμένη περίοδο διαμονής, αφού χρησιμοποιήσει κανείς την θεώρηση θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να πάρει παράταση υπό συγκεκριμένε προϋποθέσεις. Σύμφωνη προσοχή όμως, η περίοδος αυτή, η παράταση δηλαδή, να είναι συγκεκριμένη, πεπερασμένη και να υπόκειται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Όσον αφορά τη διαδικασία, όπως προείπα, ε, να δούμε λίγο τις κατηγορίες των πιθανών δικαιούχων και συμφωνώ με τον ε, εισηγητή θέλουμε αποδείξεις ε, διαμονής σε διάφορα κάτι μέλη. Δηλαδή θέλουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, αποδείξεις ε, συγκεκριμένες. Όσον αφορά την επεξεργασία της αίτηση, το είχα πει και εγώ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, πιστεύω ότι το κράτος μέλος που πρέπει να επεξεργάζεται την αίτηση πρέπει να είναι το κράτος το οποίο θα μείνει ο ετών το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Α πούμε έρχεται κάποιος από τη Λατινική Αμερική και α πούμε ότι θα περνούν από τη Μαδρίτη. Ε, ωραία, περνούν από τη Μαδρίτη αλλά δεν θα μείνουν καθόλου εκεί. Θα κινηθούν στις ε, χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Είναι λογικό να κάνουν την αίτηση στην ε, Μαδρίτη ή είναι πιο λογικό ας πούμε αν πήγαινε στη Γερμανία να κάνουν την αίτηση στην Γερμανία και να χορηγηθεί εκεί η θεώρηση. Το σημείο εισόδου μου θυμίζει λίγο Δουβλίνο, ξέρετε. Μην τα βλέξουμε τώρα με το <laughs> Δουβλίνο, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην καταλήξουμε σε ένα ατομικό κατά περίπτωση Δουβλίνο, να θέσουμε ένα διαφορετικό κανόνα εδώ. Έχω τις επιφυλάξει μου επίσης όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες. Και σε αυτό δεν τις βλέπουν καλό μάτι αντιλαμβάνομαι. Άλλωστε δεν μπορούν να υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες. Εγώ πιστεύω ότι αν θεσπίσουμε ένα γενικό σύστημα που τα καλύπτει όλα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αποκατασταθούν καλές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, τότε αυτό το σύστημα νομίζω καλύπτει τους πάντες με τρόπο ικανοποιητικό. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά τις ε, θεωρίες περιήγησης. Θα ξαναδιαβάσω τη σημεία μου και ίσως <laughs> ξεκαθαρίσω τι ήθελα να πω, αλλά όπως είπα συγγνώμη καθυστέρησα, άργησα και δεν πρόλαβα να θυμηθώ τι ακριβώς θέλω να πω. Κύριε Πελερό Er. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι συμφωνώ με τις ανησυχίες του κυρίου Λόπες Αγγιλάρ για το πού κατευθύνεται η πρόταση. Εγώ πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν ήταν μια καλή πρόταση βασιζόταν ε, στα πλεονεκτήματα του να έχουμε ένα πιο εύκολο σύστημα για τους ανθρώπους που παρνούν συχνά τα σύνορα και που ταξιδεύουν σε μία σειρά χωρών στην Ευρώπη. Ουσιαστικά θέλαμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Όμως, ε, από ό,τι φαίνεται τώρα, ο εισηγητής έχει επικεντρωθεί στα μειονεκτήματα παρά στα πλεονεκτήματα. Επομένως, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηρίξω την πρόταση του εισηγητή. Θα πρέπει να καταθέσουμε μια σειρά τροπολογιών. Φυσικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβασμό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω τίποτα που μπορώ να υποστηρίξω στην πρόταση του εισηγητή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Μπουσίετ. Κυρία Βερσιά, σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που έφτασα καθυστερημένα. Μικρόφωνο παρακαλούμε για την ομιλήτρια. Δυστυχώς δεν είχα χρόνο να εξετάσω λεπτομερώς την πρόταση του κυρίου Ορτφέ γιατί έφτασε καθυστερημένα. Απλώς ε, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Γκιλέρ και την κυρία Σεμπέλου. Εγώ πίστευα ότι η λογική που έπρεπε να ακολουθήσουμε εδώ ήταν της απλούστευσης ε, και για τους δικαιούχους αλλά και για τις υπηρεσίες μας ε, στο εξωτερικό και νομίζω ότι οι προτάσεις του κυρίου Ορτφέ ακριβώς οδεύουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ίσως λοιπόν να μην έχουν προσδιοριστεί καλά οι δικαιούχοι, να το σκεφτούμε. Εγώ νομίζω ότι τι διακυβεύεται εδώ, είμαστε υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του χώρου Σέγγεν και επισκευόμαστε ή όχι το χώρο Σέγγεν ε, και νομίζω ότι κατάλαβα τι σκέφτεται ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των διμερών συμφωνιών και των θεωρήσεων που εκδίδονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τελικά με ποια λογική συμφωνούμε. Είτε συμφωνούμε με τη μία λογική είτε με την άλλη λογική. Άκουσα τι είπε και ο κύριος Ντεπρέ όταν ε, αναφέρθηκε στο Δουβλίνο. Πραγματικά νομίζω ότι με το Δουβλίνο ακριβώς αυτό που δεν λειτουργεί είναι ότι ε, δεν ακολουθεί μια ευρωπαϊκή λογική η πρόταση. Χρειαζόμαστε περισσότερη λογική και ελληνική στο χώρο Σέγγεν και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και νομίζω ότι όλα αυτά πήγαιναν προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι περιορισμοί των θεωρήσεων αντίκειται στη βούληση που έχουν εκφράσει διάφορα θεσμοί και φυσικά από το Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν αλλά και κάποια κρατημέλη όταν ε, είπαν ότι ήθελαν να προσελκύσουν ε, νέους πτυχιούχους, ε, εγκεφάλους και φυσικά όταν δεν προωθούμε αυτά τα μέτρα προκαλούμε ακριβώς το αντίθετο και αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία κυρίως σχετικά με τους νέους που προσπαθούν ε, να σπουδάσουν ε, και να βρουν απασχόληση, δυστυχώς ε, όλο και περισσότερο απομακρύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μπλε κάρτα δεν είναι επιτυχής. Αν δεν αλλάξουμε λογική θα συνεχίσουμε να έχουμε αποτελέσματα διαφορετικά από αυτά που επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Στίβενς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για το θέμα της α, βίζας για ανθρωπιστικούς λόγους, Θα ήθελα να αναφερθώ στα δύο σημεία από κοινού το προηγούμενο και αυτό που συζητούμε τώρα. Χαίρομαι που ο εισηγητής συμφώνησε ότι αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και όλους αυτούς οι οποίοι ε, ζητούν διεθνή προστασία. Θεωρώ ότι βεβαίως ε, αναφερόμαστε σε άτομα τα οποία εγκαταλείπουν τις χώρες τους στις οποίες απειλούνται οι ζωές τους. Και αναρωτιέμαι αν ε, υπάρχει μία πρόβλεψη. Εδώ απλώς ε, προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να ελέγξουμε όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με έναν ε, τρόπο οργανωμένο και εγκαίρος. Καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι αυτή η βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους πρέπει να είναι κάτι το τελείως ξεχωριστό το θέμα των θεωρήσεων που δίνονται για τις χώρες Σέγγεν δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τις ε, ανθρωπικές βίζες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κιούμπερ, ευχαριστώ πολύ. Άργησα γιατί ήμουν ε, με τον Υπουργό από τη Σουηδία που επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει το σημείο 17. Τότε θα περάσω το 18. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, τους πολυάριθμους πρόσφυγες, και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, θα αντιμετωπιστεί με το περαιτέρω άνοιγμα των συνόρων μας. Βλέπουμε την ανεργία των νέων στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, στην Ελλάδα. Τι θα κάνουμε, θα επιτρέψουμε ακόμα περισσότερους ξένους να μπουν στην Ευρώπη και να πάρουν τις δουλειές των νέων Ευρωπαίων. Υπάρχουν προβλήματα στον έλεγχο στα σύνορα. Μα τι προσπαθεί να κάνει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν φτάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη και τους επιτρέπουμε να διαμείνουν για κάποιες μέρες, για κάποιους μήνες. Με ποιο τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε αν πραγματικά θα τηρήσουν αυτές τις ε, ημερομηνίες που τους δίνουμε για να εγκαταλείψουν την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μαύρη εργασία. Δεν καταλαβαίνω τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Η θεώρηση περιήγησης επίσης ε, θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Τζάι του Οκτωβρίου ε, προκειμένου να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επιτυχύνουμε τις εργασίες. Θα έχουμε μια συζήτηση ανατολισμό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και όσους πήραν το λόγο για την πρόσθεση της Κομισιόν για τη θεώρηση περιήγησης. Η Κομισιόν ε, καλωσορίζει τόσο όσα σε σχέση με την ανάγκη εξέβρεση ε, λύση ε, για ορισμένου ταξιδιώτε που έχουν νόμο συμφέρον να ταξιδεύσουν στο χώρο Σέγγελ. Η Κομισιόν έχει καταθέσει μια ισορροπημένη πρόταση για να καλύψει αυτά τα νομικά κενά και ε, θέλουμε εδώ να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη. Εδώ στον οικονομικό αντίκτυπο δίνουμε ορισμένα αριθμητικά στοιχεία που συνοδεύουν την πρόταση και έχουμε λάβει υπόψη ότι ο κάτοχος μιας τέτοια θεώρησης ε, θα μείνει τουλάχιστον για 91 ημέρες στο χώρο και επομένως ε, θα υπάρξει ανάπτυξη γιατί θα ταπανίσει ο άνθρωπος αυτός ε, για τη στέγασή του κτλ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι λογικά τα αριθμητικά στοιχεία που δίνουμε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνιστόσα, αλλά επίσης ε, τίθενται και πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια που πρέπει να πληρούνται. Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά τα μέσα διαβίωσης, ε, θέλουμε ακριβώς αποδείξεις για να ελεγχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο λαθρομετανάστευσης και η έλεγχη ε, ασφάλειας ισχύουν για τις θεωρήσεις Schengen, θα ισχύουν και για τη θεώρηση αυτή Πρόκειται λοιπόν για μια ισορροπημένη πρόταση και οι ανησυχίες σε ό,τι αφορά την παράνομη μετανάστευση έχουν ληφθεί υπόψη. Σε ό,τι αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογή της πρότασης, η Κομισιόν θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογή που προτείνει ο είναι πολύ στενό περιορίζεται στο επαγγελματικό ενδιαφέρον, πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και σε ορισμένε περιπτώσεις θα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υλοποιηθεί παραδείγματος χάρη σε σχέση με τους αθλητές ή ορισμένους καλλιτέχνες που κάνουν εμφανίσεις ζωντανέ. Οι προτινόμενες τροπολογίες αφήνουν εκτός άλλες κατηγορίες ανθρώπων που μπορεί να έχουν νόμιμο συμφέρον να μείνουν πάνω από 90 μέρες στο χώρο Σέγγεν, χωρί να μένουν ε, σε ένα μόνο μέλο, μέλος, το χάρη με μονομένοι ταξιδιώτε, ε, τουρίστε, συνταξιούχοι. Ορισμένοι που δεν υπόκειται στην απέτηση θεώρηση, το χάρη, και που ε, θα έφτανε ελάχιστο κίνδυνο ασφάλεια, να γνωρίζετε στο σχέδιο έκθεση και σχετίζεται και με το θέμα των διμερών συμφωνιών η Κομισιόν έχει πει ότι δεν είναι συμβατέ με τι διατάξει τη συνθήκη για μια κοινή πολιτική θεωρήσεων, δημιουργούν ε, ανασφάλεια δικαίου και θέτουν προβλήματα και στους ταξιδιώτες αλλά και στους και σε σχέση με το πόσο πρέπει να διαρκεί η παραμονή στο χώρο Σέγγεν δεν υπάρχει διαφάνεια. Επίση, η Κομισιόν δεν έχει προτείνει καταγγελία αυτών των δημοσιογραφιών θα συνεχίσουν να ισχύουν γιατί μπορεί να καλύπτουν άλλα ζητήματα, αλλά θέλουμε απλώ να τι ευθυγραμμίσουμε με τους κανόνες του κεκτημένου Σέγγεν σχετικά με τη διάρκεια παραμονής στο χώρο Σέγγεν, δηλαδή 90 μέρες σε μια περίοδο 180 ημερών. Θέλουμε απλώ να έχουμε κοινού κανόνε για όλου του υπηκόους τρίτων χωρών. Έχουμε μια μεταβατική περίοδο που δίνεται και πιστεύουμε ότι με αυτό δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι το κατάλληλο νομοθέτημα για να λύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στην πράξη. Τώρα για τα συνοδευτικά έγγραφα, η Κομισιόν ήδη είχε προτείνει πρόσθετα έγγραφο που πρέπει να παρουσιάζει, να καταθέτει ο ετών σε ό,τι αφορά τα μέση διαβίωσης, παραδείγματο χάρη. Θα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις για όλη την περίοδο της σκοπουμένης παραμονής και θεωρούμε ότι τα πρόσθετα έγγραφα που απαιτούνται είναι επαρκή σε ό,τι αφορά τώρα τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κρατημέλη. Είναι ενδιαφέρουσα η, η πρόταση αυτή. Η Κομισιόν επί της αρχής δεν είναι αντίθετη. Ε, η διαβούλευση αυτή θα πρέπει να γίνεται μέσα σε μια λογική περίοδο. 30 μέρες μπορεί να είναι μια μεγάλη προθεσμία, όμως ε, θα συνεχίσουν να ισχύουν και διατάξεις για την ε, πρώτερη διαβούλευση. Υπάρχει μια νέα πρόταση για τον ορισμό ενός του οργανωτή organizer. Αυτό δεν θα ισχύει για ορισμένε κατηγορίε ετούντων που προτείνει η Κομισιόν, πριν του χάρη μονομένου ταξιδιώτε. Και το ίδιο ισχύει και για τι τροπολογίε για το αρμόδιο κράτο μέλο. Είναι ενδιαφέρουσε οι τροπολογίε αυτέ και νομίζω ότι αυτό και είναι ένα θέμα που τέθηκε και από άλλου βουλευτέ. Η Κομισιόν ευχαρίστω να το διερευνήσει και θα πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό για αυτά τα αρμόδια κρατημέλη. Το ίδιο ισχύει και για τους όρους παράτασης. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το επιλύσουμε. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τη διάταξη που προτείνει ο εισηγητής, ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να συνδυαστεί η θεώρηση περιήγησης με άλλα είδη ε, θεωρήσεων ή με άδειες διαμονής. Φαίνεται μια λογική πρόταση Αυτά είναι λοιπόν κάποια σύντομα σχόλια για το σχέδιο έκτασης και πάλι ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δουλειά του επί της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ. Ο, λίγος, ο λόγος του κύριου Χτεφέ για κάποια καταλητικά σχόλια. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους και όλες για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, ακόμα και τις ερωτήσεις, τις αντιρρήσεις που συμπληρώνουν αυτή τη διαβούλευση επί της συγκεκριμένης Δεν έχουμε χρόνο να απαντήσω με λεπτομέρειες ε, εφ' τη της Μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζήτηση σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Ε, θα τα ξαναπουμε ουτω ούτως ή άλλως μεταξύ συγητών. Δύο-τρία πράγματα όμω. Ο κ. Αγγιλάρ είπε ε, δικαίως ότι υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, οι τουρίστες. Τα κράτη-μέλη επέμειναν ως προς το εξής. Υπάρχουν κίνδυνοι κατάχρησης, απάτης, κίνδυνος ασφάλειας, κίνδυνος παρατυπής μετανάστευσης θέματα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα. Και είναι δύσκολο ε, προκειμένου να υποβάλει κανεί ε, έγγραφα τα οποία να παρέχουν 100% ασφάλεια. Για να καθησυχάσουμε λοιπόν τα περισσότερα κάτι κράτη-μέλη. Τα κάτι μελη αυτά έχουν φόβου, του οποίου λοιπόν συμμερίζομαι. Θα ήμουν υπέρ τη σύνεση εδώ. Δηλαδή, να προσδιορίσουμε κατηγορίες πολύ συγκεκριμένες και όχι όπως να δούμε πώς θα γίνει και μετά από δύο χρόνια και πώς πήγαμε κλπ. Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε περιορισμένα μαζεμένα στην αρχή και μετά να επεκταθούμε και όχι το αντίθετο. Τώρα για τους ερευνητές, είπε ο κ. Αγγιλάρ, και τους αφηρητές ε, ε, πείτε μου όμως, κύριε Αγγιλάρ, ε, κάτι πολύ βασικό, τι θέλουμε να πετύχουμε εδώ. Ποιος είναι ο στόχος. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια θεώρηση η οποία θα ανταγωνίζεται άλλες κατηγορίες θεωρήσεων. Και το πράγμα το οποίο θα οδηγήσει αναγκαστικά σε σύγχυση της ε, προξενικής υπηρεσίας. Ή θέλουμε να δημιουργήσουμε μια θεώρηση, η οποία απλώ θα διευκολύνει συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων που μεταβαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη. Σε αυτό να επικεντρωθούμε λοιπόν. Πολύ συγκεκριμένε κατηγορίε με πολυ τη σαφήνεια Αυτές δηλαδή τις κατηγορίες που θέλουμε να διευκολύνουμε επειδή ακριβώ μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη. Ο Ζεράν Ντεπρέ έθεσε διάφορα θέματα. Τους φοιτητέ, τη διάρκεια ισχύω. το ποιο κράτος ήταν υπεύθυνο για την επεξεργασία τη αίτης κλπ. Και, είπε κάτι με το οποίο συμφωνώ. Τώρα όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες. Πιστεύω ότι η Κομισιόν πρέπει να οργανώσει συζητήσεις με τα τη μέλη σε άλλο χώρο όμως, σε άλλο πλαίσιο, όχι εδώ σήμερα. Όπως είπε του Ζεράρ, δεν ξέρουμε πόσες τέτοιες συμφωνίες υφίστανται καταρχά. Δεν ξέρουμε ποιες χώρε εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών. Ούτε γνωρίζουμε τι επιπτώσει, στην περίπτωση που ληφθεί μία μονομερής απόφαση στο πλαίσιο ενό κανονισμού. Εξού και η θέση μου, την οποία εξήγησα προηγουμένως. Κύριε Τόμασιτ, αναφέρθηκε στα προβλήματα ασφάλειας, ανησυχεί, συμμερίζουμε τι ανησυχίες τη, συμμερίζουμε την αλυσή της. Κύριε Βαλερό, αναφέρθηκε σε κάποια άλλη λογική, η οποία κατά την τοπική άποψη είναι εντελώ διαφορετική. Ε, δεν έχω κάποιο άλλο σχόλιο, δεν πιστεύω ότι διαφωνούμε. Αυτά λοιπόν εντάχει. Αυτά είναι τα θέματα που θέλησα να σχολιάσω. Από εκεί πέρα στη διάθεση των συναδέλφων για να το ξανασυζητήσουμε στην μεγαλύτερη βάθος αν χρειαστεί. Πρόεδρος, Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών είναι 25 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. 25 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Όπως και την προηγούμενη πρόταση για τον κώδικα θεωρήσεων. Ε, είμαστε λίγο πιο μπροστά από το πρόγραμμα, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Παρουσίαση από τον ε, διευθυντή τη Ιουλίζα, τον κύριο Κρουμ Γκάρκοφ. Καλό τον κύριο Γκάρκοφ. Εδώ, δίπλα μου για την παρουσίασή του. Okay. Okay. Then... Πολύ ωραία. Από τη συνάδελφη, όπως γνωρίζετε, οι εργασίε για την νομοθετική πρόταση όσον αφορά το πακέτο για τα έξυπνα σύνορα έχουν ανασταλεί. Αποφασίστηκε να εκπονήσουμε μια επιπλέον τεχνική μελέτη, κάτι το οποίο συζήτησαμε ήδη στην Επιτροπή αυτή, και από εκεί πέρα να περάσουμε σε μια φάση πρακτικών δοκιμών από την Ιουλίσσα. Οι δοκιμέ αυτέ συνεχίζονται, είναι εξελίξη, και οι συγητέ μα είχαν την ευκαιρία να τα δουν όλα αυτά στην πράξη στην Φιλανδία. Τον Ιούλιο με την ε, ενδιαμεσή έκθεση για τις δοκιμές αυτές και αυτό ακριβώ το κείμενο, αυτά τα αποτελέσματα θα μας παρουσιάσει ο κ. Γκάρκοφ σήμερα. Δίνω τον λόγο στον κύριο Γκάρκοφ και αμέσω μετά θα μιλήσουν οι φοιητές και οι άλλοι βουλευτές. Κύριε Γκάρκοφ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Όπως πάντα χαίρομαι που σας ξαναβλέπω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για να σας ενημερώσω περί της πρόοδου στον σημαντικό αυτόν τομέα, το πιλωτικό έργο στον τομέα έξυπνα σύνορα. Νομίζω ότι έχουμε φέρει και κάποιες διαφάνειες, δεν ξέρω αν μπορούμε να τις δούμε. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα Τα βλέπουμε όμως. Λοιπόν, να σας ενημερώσω για το πιλωτικό έργο. Να θυμίσω το γενικότερο πλαίσιο, τι σημαίνει έξυπνα σύνορα και τι σημαίνει ε, το συγκεκριμένο πιλωτικό έργο. Το επόμενο παρακαλώ. Είδαμε μια γενική εικόνα των εξωτερικών μας συνόρων. Υπενθυμίζω ότι έχουμε πάνω από 7.000 χιλιόμετρα χερσών συνόρων και πάνω από 42.000 χιλιόμετρα θαλασσίων συνόρων. Σημεία διέλευσης 1.800 από τα οποία παίρνουν κάθε χρόνο 700 εκατομμύρια άνθρωποι. Έχουμε 700 εκατομμύρια διελεύσεις το χρόνο. 30% αυτών των διελεύσεων αφορούν υπηκούς τρίτων χωρών. Και αυτά τα νούμερα αναμένεται να διπλασιαστούν πολύ σύντομα. Με άλλα λόγια, η ζήτηση ούτως υπήρχε στα εξωτερικά σύνορα αυξάνεται. Το οποίο σημαίνει χρειαζόμαστε περισσότερους συνοριοφύλακες ή πρέπει να βρούμε εξυπνότερους τρόπου, τρόπους δηλαδή την σύγχρονη τεχνολογία για να καταστήσουμε την διαχείριση των συνόρων πιο έξυπνη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η πρωτοβουλία έξυπνη διαχείριση συνόρων έχει θετικέ επιπτώσει σε τρει τομεί. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Πρώτον, όσον αφορά την διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι άνθρωποι θα διέρχονται ευκολότερα τα σύνορα. Την, την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Πρώτον, διευκόλυνση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών ευκολότερη διέλευση λοιπόν των εξωτερικών συνόρων, πιο αποτελεσματική και αποδοτική συνορική εκεί έλεγχη και εξίσου σημαντικό, αν όχι πιο σημαντικό, προστασία της εσωτερικής ασφάλειας. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας έξυπνη διαχείρισης συνόρων. Να θυμίσω σε τι συνίσταται το πιλωτικό έργο. και μετά θα σας πω και μερικές ε, λεπτομέρειες παραπάνω. Λοιπόν, το πιλωτικό έργο, με δύο λόγια, σύντομη επισκόπηση, πρόκειται για μια ευρεία εφαρμογή πρωτοβουλία, μικρή όμω διάρκεια, καταλαβαίνει σχεδόν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 11 κράτη-μέλη υποστηρίζουν το έργο αυτό και 10, σε 17 σημεία εισόδου. Ο λόγος είναι απλός. Χρειαστήκαμε ένα πλειοτικό έργο για να δοκιμάσουμε διαφορετικά σενάρια, διαφορετικές τεχνολογίες και στους τρεις τύπους συνόρων. Ενέργεια σύνορα, χερσαία και θαλάσσια. Έτσι ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες ολοκληρωμένες συστάσεις σχετικά με το ποια είναι η καλύτερη τεχνολογία, ποια είναι η καλύτερη μέθοδος να πετύχουμε τους στόχους της πρωτοβουλίας. Χρονοδιάγραμμα. Οι προετοιμασίε για το πιλωτικό ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2014. Ολοκληρώσαμε τι προετοιμασίε τον Φεβρουάριο και πέρασαμε στην φάση της εκτέλεσης, της υλοποίησης, τον Μάρτιο του 2015. Κοντεύουμε να κλείσουμε το έργο, να το ολοκληρώσουμε και η υποβολή εκθέσεων θα γίνει από τον Οκτώβριο στον Νοέμβριο του 2015. Η έκθεση υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της συμφωνίας που υπεγράφει ε, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αντικείμενο. 109 συγκεκριμένες ερωτήσεις, 13 ε, σύνθετες υποθέσεις βάση τα ερωτήματα που έθεσε η Κομισιόν το 2014. Και έχουμε και τις μελέτες ε, που έγιναν όχι επί τόπου αλλά στο γραφείο από τις υπηρεσίες υποστήριξη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Διαδικασίες, ε, εναλλακτικέ διαδικασίες στην περίπτωση που το σύστημα καταρρεύσει παράδειγμα. Τι γίνεται στην περίπτωση λοιπόν χ ε, διακινητών με ψί διακινημένου κλπ. Όλα αυτά είναι εν εξελίξη όπως είπα. Το αποτέλεσμα των διαφόρων δοκιμών αλλά και των μελετών θα ενσωματωθούν σε μια τελική έκθεση. Τονίζω επίση το γεγονό ότι επιπλέον των τεχνικών πτυχών του έργου αυτού συνεργαζόμαστε με τις αρχές που ασχολούνται που εμπλέκονται στα δικαιώματα του ανθρώπου. Ε, στην τελική λοιπόν έκθεση θα έχουμε και τις απόψεις ε, του οργανισμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου, των θεμελιδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πού βρισκόμαστε λοιπόν. Ε, αν και εγώ ασχολούμαι καθημερινά με την υλοποίηση, όπως είπα τελειώνουμε σε λίγο Βάση του χρονοδιαγράμματος. Τέλη Σεπτεμβρίου λοιπόν θα είμαστε έτοιμοι. Να τονίσω με την ευκαιρία ότι, όπως είπα, κινούμεθα βάση του χρονοδιαγράμματος, δεν έχουμε καθυστερήσει, παρά τις τεχνικές δυσκολίες, τις προκλήσεις, γενικά όμως ο οργανισμός και το προσωπικό συνεργάστηκαν ικανοποιητικά. Πάμε πολύ καλά και να μένουμε να ολοκληρωθεί η υλοποίηση βάση του αρχικού χρονοδιαγράμματος εντός προθεσμίας η έκθεση το ίδιο. Η ενδιάμεση έκθεση με την ευκαιρία υπευλήθη εγκαίρως. Διαβάσαμε και μερικά ενδιαφέροντα ευρήματα όσον αφορά τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έξυπνη διαχείριση. Τι μένει ακόμη τώρα, ε, όπως είπα, θα βάση χρονοδιαγράμματος, χωρίς καθυστέρηση. Ε, να σας πω τώρα τις κατατόπους εξελίξεις. Διάφορα κράτη-μέλη συμμετέχουν, σε 17 σημεία εισόδου, σημεία διέλευσης. Εδώ βλέπετε για τα ενέργεια σύνορα τελειώσαμε ήδη στο, στη Φραγκφούρτη και στο Φραλντεγκόλ στο Παρίσι. Τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε τα αποτελέσματα και κλείνουμε με τα ενέργεια σύνορα. Όσον αφορά τα χερσαία σύνορα, συνεχίζονται οι δοκιμές σε διάφορα σημεία διέλευσης. Έχουμε όμως και εκεί προχωρήσει πολύ. Το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων έχουν καταγραφεί και εδώ δεν έχουμε καθυστερήσει καθόλου και στα θαλάσσια σύνορα τώρα έχουμε συγκεκριμένε περιπτώσεις που αφορούν ε, χρήση της τεχνολογίας σε κινούμενα τρένα ή οι επιβάτες σε αυτοκίνητα όσον αφορά τις τοποθεσίες λοιπόν και εδώ πηγαίνουμε καλά. Εδώ βλέπετε την πρόοδο ανά φάκελο, ανά τύπο δοκιμής. Έχουμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο γιατί αυτά είναι τα στοιχεία τέλους Αυγούστου, δηλαδή τα ποσοστά έχουν ανέβει ακόμη περισσότερο. Το 70 ας πούμε 80 ήδη και ούτω καθεξής. Άρα και εδώ θα τηρήσουμε την υποθεσμία. Αν και πρόκειται για προκαταρκτικά αποτελέσματα, ήδη πρέπει να σας πω έχουμε στα χέρια μας πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Στην ενδιάμεση λοιπόν έκθεση που κατήρθησε ο οργανισμός μέσα Ιουλίου, όπως ε, προείπα, υπάρχουν ευρήματα τα οποία δείχνουν προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Σχετικά δηλαδή με, τις, με τη συνεισφορά της τεχνολογίας στη διαχείριση των σημείων διέλευσης. Τονίζω ότι Υπάρχει ευρεία αποδοχή αυτών των νέων μεθόδων και από τους επιβάτες, τους ταξιδιώτες και από τους συνοριοφύλακες. Και τούτο, διότι σύμφωνα με την διαμεσή έκθεση και τα σχετικά στοιχεία, το πλήθος των ε, συμμετεχόντων ήταν θετικό σε το πάνω από 90%. Όσον αφορά τους συνοριοφύλακες, σε διάφορες τοποθεσίες, και εκεί είχαμε μια πολύ θετική υποδοχή του νέου συστήματος, των νέων τεχνολογιών. Κάτι άλλο, πολύ σημαντικό προγραμματικό έβριμα, το οποίο θα το επεξεργαστούμε περαιτέρω βεβαίω εν της τελικής έκθεσης, είναι η αξιοπιστία της χρήσης βιομητρικών δεδομένων και του σχετικού εξοπλισμού, που κάνει δηλαδή, τις διαδικασίες πιο αποτελεσματικές. Από τα προκαταρκτικά στοιχεία φέρεται σαφώς ότι για την επαλήθευση χαρακτηριστικών του προσώπου, δακτυλοσκόπηση κλπ. Δεν χρειάζεται και πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με τις σημερινέ διαδικασίες. Από την άλλη μεριά όμως εννοείται έχουμε πολύ ψηλότερη αξιοπιστία και ασφάλεια. Άρα λοιπόν θετικός εν τέλει ο αντίκτυπος τόσο για τους ταξιδιώτες αλλά και για τους νοριοφύλακες. Και αυτό θα το επεξεργαστούμε περαιτέρω, θα μαζέψουμε όλα τα στοιχεία και θα διατυπώσουμε φυσικά εν συνεχεία συστάσεις και προτάσεις. Η αξία του πιλωτικού έργου δεν είναι μόνο να μας βοηθήσει να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με το ποια είναι η βέλτιστη μέθοδος, αλλά να δούμε και που υπάρχουν προβλήματα υλοποίηση για να πετύχουμε ε, τον αρχικό στόχο. Αυτά είναι μερικά από τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία συμπεριλήφθησαν στην προκαταρκτική, στην διάμεση έκθεση. Πρώτον, για τον οργανισμό είναι σαφές ότι κάποιες διαδικασίες ε, ελέγχου συνόρων, ε, ας πούμε η δακτυλοσκόπηση σε ένα τρένο που κινείται ή η δακτυλοσκόπηση επιβατών αυτοκινήτου κλπ. Εκεί ε, ενδεχομένω δεν έχουμε καταλήξει, δεν έχουμε στα χέρια μα αρκετή τεχνολογία, ικανή τεχνολογία. Θα το γράψουμε αυτό στην τελική έκθεση, είναι σημαντικό έβριμα, αλλά όπως είπα, λίγο πολύ έχουμε μια εικόνα των υφισταμένων τεχνολογιών που μπορούν να μας βοηθήσουν, ως κάποιο σημείο βέβαια, για να βρούμε λύσεις σήμερα και αύριο. Λοιπόν, η διαφάνεια, να μην επισέλθουμε τώρα στα πολύ τεχνικά, όμως η ενδιαμεσή έκθεση, όπω είπα, περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα, αλλά και λεπτομέρειε λοιπόν, πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα. Πρώτον, το πιλωτικό ολοκληρώνεται τέλη Σεπτεμβρίου. Από εκεί πέρα οι ανεξάρτητες μελέτες θα συμπληρώσουν το πιλωτικό, θα ολοκληρωθούν και αυτές μέσα Οκτωβρίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν προχωρήσει πολύ αυτές οι μελέτες, αλλά όπως είπα πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουν να καταλήξουν μέσα Οκτωβρίου και θα ενσωματωθούν στην τελική έκθεση. Παράλληλα, ο οργανισμός προετοιμάζει την σύνταξη της τελικής έκθεσης που και αυτή θα έρθει στην ώρα της, τέλη Νοεμβρίου. Μια έκθεση που ευελπιστώ ότι θα μας δώσει μια έγκυρη άποψη για τις τεχνολογίες και το πώς μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των συνόρων. Είναι μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει και βάση για μελλοντικές παρομοίες προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Εννοείται για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας σε αυτήν την έκθεση. Εμείς έχουμε ορίσει δύο συγητές, Δίας Δεμέρα και Παϊόν. Η δεύτερη συγγήτρια δεν είναι σήμερα εδώ. Θα αντικατασταθεί από την κυρία Σίπερ. Θα δώσω το λόγο όμως πρώτα στον κύριο Τίας Δεμέρα, τον πρώτο συγητή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν μιλήσω για την αξιολόγηση της ενδιάμεσης έκθεσης που μας παρουσίασε ο κ. Γκάκοφ. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ και η κυρία Φαγιόν ότι είμαστε δυσαρεστημένοι γιατί θεωρούμε ότι η Κομισιόν προέβη σε μια κακή πρακτική και για μια ακόμη φορά διακυβεύεται το πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας. Και δυστυχώς αυτό έχει συμβεί πολλάκις. και ουσιαστικά αμφισβητεί το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Στις 26 Ιουνίου, όπως φαίνεται, όλα αυτά τα ξέρουμε ανεπίσημα, αλλά ισχύουν. Στις 26 Ιουνίου η Κομισιόν παρουσίασε σε μια συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Συνόρων στο Συμβούλιο ένα έγγραφο που λέγεται μη έγγραφο, ένα non-paper, επίσημο έγγραφο που μελετά τη δυνατότητα να θεσπιστεί ένα γρήγορο σύστημα και το οποίο θα έπρεπε να συμπληρώσει ίσως και να αντικαταστήσει το πρόγραμμα RTP. Και ουσιαστικά αυτή είναι η έκθεση για την οποία είναι αρμόδια η κυρία Φαγιών. Τώρα, χωρίς να μπω στην ουσία της υπόθεσης, Κανείς δεν μας κοινοποίησε επισήμως αυτό τον επίσημο έγγραφο, αυτό το non-paper και σας ήθελα να πω ότι μια τέτοια πρόταση θα είχε τεράστιο αντίκτυπο στη δέσμη μέτρων για το εφή e σύνορα. Έτσι λοιπόν, απαιτώ ως συνσηγητής και τα δύο όργανα να την χάνουν ίση μεταχείρισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει όλε τι πληροφορίε για τα θέματα που συζητούνται. Μόνο με αυτόν τον επικοδομητικό τρόπο μπορούμε να εργαστούμε για να ολοκληρώσουμε μια τόσο πολύπλοκη δέσμη μέτρων όσο αυτή των ευφυών συνόρων. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση του κ. Γκαρκόφ. Καταρχήν, ευχαριστώ τον κ. Διευθυντή για τι εξηγήσει που μα έδωσε και θα ήθελα να πω στην ε, Επιτροπή ότι είναι πολύ καλό το έργο της ε, Ιουλίσσα. Είναι άψογο. Στις επόμενες τριάσεις ε, της Επιτροπής Λίμπες θα σας εξηγήσω ε, κάποια πράγματα σε σχέση με την επίσκεψή μας στη Φιλανδία. Σήμερα θα πω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και θέλω να ευχαριστήσω τις Ολλανδικές Αρχές, τους τεχνικούς της υπηρεσίας και τα μέλη της Γραμματείας. Σε σχέση τώρα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, θα είμαι σόφρον στις παρατηρήσεις μου αναμένοντας το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι πράγματι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα σύστημα ευφυών συνόρων είναι τεχνικά εφικτό, είναι δυνατό. Η έκθεση είναι πολύ μεγάλη, έχει 180 σελίδες και μας αναφέρει τα πρώτα αποτελέσματα ε, των, ε, της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων με 4, 8 και 10, της άρρωσης της και της ε, χρήσης ε, κάποιων θυρών και ουσιαστικά πώς αυτά ενσωματώθηκαν στο σύστημα ΒΙΣ. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να τα λάβουμε υπόψη θα πρέπει να περιμένουμε τα τελικά συμπεράσματα. Ήδη μας είπαν ότι θα τα έχουμε το Νοέμβριο και ουσιαστικά πρέπει να δούμε και ποιο θα είναι το αντίκτυπο στο ταξιδιώτη. Ουσιαστικά οι χρήστες σε 190 σελίδες έχουν εκφράσει μεγάλη ικανοποίηση. Επίσης ε, βλέπουμε και ικανοποίηση από την πλευρά των συνεροφυλάκων καθώς και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές για να έχουμε κάποιες ταχύτερες διαδικασίες κατά τη διέλευση των συνόρων. Η επιτέχυνση της διέλευσης των συνόρων είναι ο κύριος στόχος και Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να υλοποιηθεί αυτή η ταχεία διέλευση των συνόρων και πρέπει να αναλύσουμε και να δούμε πώς αυτός ο στόχος μπορεί να είναι εφικτός και συμβατός με άλλους δευτερεύοντες στόχους όπως η πρόσβαση των αρχών ασφαλείας, των δυνάμεων ασφαλείας στα δεδομένα. Επίσης το θέμα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην ταχύτητα της συγκέντρωσης των στοιχείων την ποιότητα των δεδομένων και η ε, δυνατότητα χρήσης των στοιχείων αυτών. Θα σας ε, θέσω κάποιες ερωτήσεις, τέσσερις, για να απαντήσετε. Καταρχήν, ποιες είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ε, έγιναν λάθη, υπήρξαν αποτυχίες σε αυτές τις δοκιμές. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί, να τους γνωρίζουν και οι συνάδελφοι. Δεύτερον, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχαμε επιτυχία της παθητικής ταυτοποίησης. Σε σχέση τώρα με τα βιομετρικά στοιχεία από τα πρώτα στοιχεία μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι καλύτερη ή όχι η συνδυασμένη χρήση χρηση δεκτυλικων αποτυπωμάτων, της αναγνώρισης του προσώπου και της σύριδας. Και τέλος, η τελική εκδοχή για το πιλωτικό σχέδιο. Πράγματι θα μας την παραδώσετε αυτή την τελική εκδοχή το Νοέμβριο, γιατί από αυτό θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να κινηθούμε εγκαίρως ή αν θα καθυστερήσει μια νομιστική πρόταση. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σίπερ που αντικατεστα την εισηγήτρια, την κυρία Φαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν είναι εδώ η εισηγήτριά μας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να στοχεύσω κάποια από τα σημεία που πρέπει να αναφερθούν. Φαίνεται ότι είναι σε πρώτο στάδιο η πρόταση και δεν μπορούμε να φτάσουμε σε τελικά συμπεράσματα. Φαίνεται ότι μόνο κάποια από τα αναμενόμενα αποτελέσματα ουσιαστικά φαίνεται να καλύπτονται και δεν ε, εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές λίστες, δεν έχουν ελεγχθεί από τεχνολογικής απόψεως. Η κυρία Φαγιών ειδικά θα ήθελε να απαντηθούν κάποια ερωτήματα όπως πολύ συγκεκριμένα ποιες είναι οι περιπτώσεις ε, ταξιδιωτών και ε, επιβατών που χρησιμοποιήθηκαν, ποιο είναι το ποιοτικό αν θέλετε, όριο που τέθηκε. Δεν είναι καθόλου σαφές ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τέτοια ε, κατόφλια. Η χρήση θηρίδων, η... το κατά πόσο είναι ευκολόχρηστα και φιλικά προς το χρήστη αυτά τα συστήματα και βεβαίως γνωρίζουμε το πόσες προσπάθειες έχει κάνει το ΛΙΖΑ, αλλά η ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Το πιλετικό πρόγραμμα δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο. Σήμερα δεν βλέπουμε συγκεκριμένες συστάσεις να μπορούν να βγουν από αυτό το πρόγραμμα. Και θα θέλαμε να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει και ποια είναι τα ποσά τα οποία θα δαπανηθούν από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βερζά έχει ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον εισηγητή όσον αφορά ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε αρκετά υποχωρήσει όσον αφορά αυτό το θέμα όσον αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα και εκπλήσωμαι γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποια άλλα εναλλακτικά προγράμματα τα οποία όλοι γνωρίζουν εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευτυχώ που ο εισηγητής μπόρεσε να ενημερωθεί έμεσα με πλάγιο τρόπο αλλά αυτό δεν μου φαίνεται ορθό και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει η συνθήκη του Λισαβόνας όταν πρόκειται για τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί αλλού βλέπουμε να ε, εφαρμόζονται ενώ εδώ σε αυτή τη διαδικασία όχι. Χωρίς λοιπόν να αμφισβητήσω την εργασία που κάνει η ε, Λίζα, θα ήθελα να πω ότι κατά κάποιο τρόπο και εγώ Αμφισβητώ εδώ τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς ε, να ε, βγάλει από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα σε σχέση με την δική μας πρωτοβουλία. Μου φαίνεται ότι καταρχήν δεν είναι αρκετά αυτά που κάνει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα καθότι περιορίζεται στο τεχνικό μόνο θέμα ενώ δεν πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα. Χαίρομαι αν κατάλαβα τουλάχιστον καλά αυτό που είπατε, ότι ο εντοπισμός μέσω βιομετρικών στοιχείων που βασίζονται στην ήριδα είναι μια ε, εναλλακτική λύση, μια επιλογή την οποία εγκαταλείπεται, διότι δεν πιστεύω ότι αυτό το σύστημα μπορεί να είναι αξιόπιστο. Θα δούμε βεβαίω τι θα βγει από αυτήν την τεχνική μελέτη, αλλά όποιο και να είναι το αποτέλεσμά της, ο, υπάρχει θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πρόκειται για μία διαδικασία η οποία είναι πολύ παρεμβατική για τους Ευρωπαίους πολίτες. Μιλάμε επιπλέον πολύ για την δημοσιονομική ε, πειθαρχία, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Εδώ ξαφνικά για ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεπεράσει το ένα δις, το κόστος τους, ξαφνικά δεν έχουμε απολύτως κανένα ε, θέμα δημοσιονομικό. Πολύ καλύτερα θα κάναμε να δαπανούσαμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να γίνεται διάσωση προσφύγων, παραδείγματος χάρη τη θάλασσα. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα συνεχίζει να έχει λόγο ύπαρξης, βλέπω ότι αλλάζουμε τους στόχους και αναρωτιέμαι επίσης αν όλη αυτή η αμφισβήτηση, η προσέγγιση μας η καινούρια έχει ενσωματωθεί ε, σε αυτά που κάνετε και ε, γιατί δεν ενημερώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Βίξτρο, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Αυτό το θέμα το παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ σίγουρα δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις αυτού του σχεδίου. Όμως έχουμε ανησυχίε για τις τεράστιες δαπάνες και είναι πράγματι αυτά τα χρήματα που δαπανούνται αρθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και θα πρέπει να υπενθυμίσω όσα υπόθηκαν από τον κύριο Δίας Δεμέρα. Και της κυρίας Δανήφαγιον ξέρω τη θέση της. Αυτά όλα δεν μας βοηθούν. Δεν βοηθούν ούτε τους ε, συνεισηγητές και ευτυχώς που τους έχουμε σε αυτόν τον οίκο. Δόξα τω Θεώ που ο Διαζαμέρα και η κυρία Φαγιόν είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν λάβει και δεόντως υπόψη και τις ανησυχίες της δικές μας των σκιώδων συγητών. Όμως, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα ήθελα να το παρουσιάσω ως ένα κακό παράδειγμα της διοργανικής συνεργασίας. Ένα πολύ κακό παράδειγμα συνεργασίας, γιατί δεν ε, μας ενημερώσατε καταλλήλως. υπήρχε διαρροή πληροφοριών ε, και κάποιοι τις ε, μετέδωσαν και αυτός είναι ο φαύλος κύκλος της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των οργάνων. Και πρέπει να υπάρξουν κάποια διδάγματα από αυτό. Θα ήθελα να επαναλάβω δεν πιστεύω ότι κάποιος στην αίθουσα αυτή θα αφισβητούσε τις καλές προθέσεις. Όμως, τα διδάγματα που εσείς και η Κομισιόν θα πρέπει να αντλήσετε από όλο αυτό είναι ότι εμείς <laughs> τώρα πια δεν το χάφτουμε όλο αυτό. Θέλουμε πληροφορίες θέλουμε να μας δώσει πληροφορίες με ένα διαφανή τρόπο. Δεν ότι πρέπει να εργαζόμαστε βάσει πληροφοριών που είναι αντικείμενο διαρροής. Είναι απαράδεκτο. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ανησυχούμε και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που θα ήθελα να θέσω, όμως προς στιγμή στέκομαι στις καλές σας προθέσεις. Όμως σας παρακαλώ να διαβιβάσετε αυτό το πολύ σαφές μήνυμα σήμερα από αυτή την Επιτροπή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Γκάρκοφ για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον που προκαλεί η εργασία μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω καταρχήν στον κύριο Ντεμέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα Ήθελα να πω και σε εσά και στην κυρία Φαγιόν και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ ότι φυσικά θα σας δώσουμε πολύ ολοκληρωμένες, όσο πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις μπορούμε στα ερωτήματά σας. Γιατί ε, θα κάποια από τα τεστ, από τις δοκιμές αποτυχημένες. Δεν απέτυχαν οι μέχρι τώρα δοκιμές που έγιναν, αλλά κάποια από αυτά τα πειράματα ήταν πολύ συγκεκριμένα και μάλιστα οι τεχνικές, η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σας είπα, υπάρχει αν θέλετε επειδή αυτή η τεχνολογία είναι πολύ υψηλού επίπεδου και προηγμένη, δεν μπορέσαμε σε όλα τα επίπεδα να ε, συλλέξουμε τα απαραίτητα δεδομένα. Γι' αυτό και είπαμε ότι κάποια από αυτά δεν είναι επιτυχημένα ή απέτυχαν. Αλλά όταν έχουμε την τελική ε, μελέτη και όταν αναλυθούν όλα αυτά τα δεδομένα, Εκείνη τη στιγμή θα μπορέσουμε να κάνουμε τον απολογισμό και να φτάσουμε σε κάποια αξιόπιστα αποτελέσματα όσον αφορά το βαθμό επιτυχίας και αποτυχίας. Σε πολλές περιπτώσεις η υπηρεσία μας συνεργάστηκε με εκπροσώπους του κλάδου, στον τομέα της βιομετρίας και άλλους επιστημονικούς κλάδους και βεβαίως κάθε φορά προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την πιο σωστή τεχνολογία αυτή δηλαδή που ανταποκρίνεται στους στόχους αυτής της μελέτης. Έχουμε κάποια λοιπόν ε, προσωρινά αποτελέσματα και μόλις έχουμε την τελική έκθεση φυσικά και θα φτάσουμε σε κάποιους τελικούς ε, σε κάποια τελικά συμπεράσματα και αν κάποια από τα πειράματα που κάναμε, τις δοκιμές που κάναμε δεν είναι επιτυχημένα, φυσικά και θα σας ενημερώσω. Ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός για να γίνει ο βιομετρικός αυτός εντοπισμός και η ταυτοποίηση. Είδαμε ότι υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί που δεν είναι καλύτεροι ίσως από άλλους, αλλά είναι ταχύτεροι. Και επαναλαμβάνω, όταν θα έχουμε την τελική έκθεση, φυσικά και θα γίνουν επιλογές που θα βασίζονται στα πραγματικά αποτελέσματα της μελέτης. Τι δηλαδή θα πρέπει να γίνεται σε πραγματικά έξυπνα συστήματα φύλαξης των συνόρων. Δεν θέλω όμως αυτή τη στιγμή να φτάσω σε συμπεράσματα πριν έχουμε τα τελικά δεδομένα για την καλύτερη ταυτοποίηση, βιομετρική ταυτοποίηση. Φυσικά και προσπαθούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες που έχουμε δώσει και πιστεύουμε ότι στα μέσα Νοεμβρίου θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την ε, μελέτη. και να μπορούμε να συλλέξουμε τα δεδομένα αυτά με τον καλύτερο και τον ταχύτερο τρόπο βάσει των δεδομένων ε, και του συστήματος που λειτουργήσε κατά τη διάρκεια του πιλωτικού προγράμματος. Ακούστηκαν και κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την επένδυση και το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Είμαι σίγουρος ότι στην τελική έκθεση θα έχετε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα όσον αφορά και τις δυνατότητες τις τεχνολογικές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχει βεβαίως μια καλύτερη χρήση τους, πιο φιλική και σε πιο αποτελεσματικές και γρήγορες διαδικασίες. Τώρα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος βεβαίως δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Και προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση αυτών των κονδυλίων από την αρχή όταν ξεκινήσαμε στις συζητήσεις μας τα κρατημέλη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ σαφές ότι αυτό που αρχικά είχαμε στοχεύσει φυσικά ξεπερνά τα ποσά τα οποία έχουν μέχρι τώρα διατεθεί. Μέχρι τώρα λοιπόν, σας λέω περίπου τα νούμερα, οι δαπάνες μέχρι τώρα είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τις δαπάνες του προγράμματος αλλά και της δαπάνες της υπηρεσίας. Τώρα, όσον αφορά τη νέα πρόταση της Επιτροπής Fast Lane για όλους, μια γρήγορη δηλαδή ταχύτητα διαδικασία, η απάντησή μου είναι όχι καθότι στα πλαίσια αυτού του πιλωτικού προγράμματος δεν είχε υποβληθεί αυτή η πρόταση. Και βεβαίως ε, μετά τη διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεχομένως αυτή η πρόταση μπορεί να εξεταστεί και να ενσωματωθεί. Προς το παρόν πάντως δεν έχει ενσωματωθεί στο πιλωτικό πρόγραμμα. Τέλος, Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, δεν επαναλαμβάνω για το κόστος, αλλά πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί η έκθεση θα δοθούν στοιχεία αξιόπιστα και για τους στόχους και για την αποτελεσματικότητα ε, αυτών, αυτού του συστήματος έξυπνων συνόρων όταν αυτό ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Θα ήθελα να στραφώ στην κύριο Ρόζεμπερκ από την Κομισιόν να μας ενημερώσει σε σχέση με τις νέες νομοθετικές προτάσεις. Το κύριο Ρόζεμπερκ, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας με τον τρόπο που εφαρμόζεται το πιλωτικό πρόγραμμα από την Ιουλίσα Πιστεύουμε ότι υλοποιείται με ένα πολύ επαγγελματικό τρόπο εντός του χρονοδιαγράμματος και με όλο το συντονισμό που απαιτείται. Και μέχρι τώρα τα αποτελέσματα έχουν ε, παραδοθεί με έναν τρόπο πολύ χρήσιμο και εγκαίρος. Ε, και τα προσωρινά συμπεράσματα που ανέφερε ο κ. Κάρκοφ ήδη μας βοηθούν για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και στην Κομισιόν και εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Μου ζητήσατε να κάνω μια ενημέρωση για το που βρισκόμαστε στη διαδικασία. Η τελευταία φορά που μιλήσαμε για τα φύση σύνορα στο Κοινοβούλιο ήταν στις 9 Ιουνίου, στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, όπου ο Επίτροπος Αβραμόπουλος μίλησε και αναφέρεται τους στόχους ε, της αναφερμένης πρότασης και τα στοιχεία από αξιολογή κομισιών για την προετοιμασία των νέων προτάσεων. Είπα ότι θα παρουσιαστούν στους συνομοθέτες στις αρχές του 2016. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι Υπουργοί Εσωτερικών συζητούν ποιες απαντήσει ε, θα δοθούν στην κρίση των προσφύγων και ως ένα μέρος αυτής της απάντησης είναι προτάσεις ε, για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ε, οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να προσχεστούν μέσα το τέλη του 2015. Αυτό λοιπόν που έχουμε κατά νου είναι ένα σύνολο συμπρασμάτων του Συμβουλίου που θα καλεί την Κομισιόν να παρουσιάσει προτάσει για την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης μέχρι τα τέλη του 2015. Αυτό το πακέτο συνήθω συμπεριλαμβάνει και προτάσεις για τα ΦΥΙ, θα πρέπει καταρχήν να δούμε αν θα αυτό θα επιβεβαιωθεί και πώς ε, αυτό θα λάβει μορφή και σε πρακτικό επίπεδο. Τι είναι εφικτό, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε και τα πορίσματα του Υγιού αλλά υπάρχει και μια δυνατότητα, μια πιθανότητα ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε την παρουσίαση της πρότασης των ευφυών συνόρων και να την καταστήσουμε διαθέσιμη πριν τα τέλη του έτους. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο σε σχέση με τον Ιούνιο όταν ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στις αρχές του 2016. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα τώρα, τι θα υπάρχει στις προτάσεις αυτές. Ξέρετε, και έχετε δει το χαρτιπορία πορείας της μελέτης αντικτύπου που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο και έχει διατεθεί για σχόλια από τον Ιούνιο και θα έχετε δει ότι οι προτάσεις ε, επικεντρώνονται σε πέντε μεγάλα ζητήματα. Το ένα είναι το θέμα της αρχιτεκτονικής, του μελλοντικού συστήματος, το δεύτερο τα βιομετρικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν και σήμερα ακούσαμε κάποια ενδεικτικά στοιχεία. Έχουμε, ε, δεν είναι πολύ πιθανό να κερδίσουν τα 10 δακτυλικά αποτυπώματα γιατί μόνο θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, μόνο θα χρειαστούμε κάτι πιο ελαφρύ. Το τρίτο θέμα αφορά τη διευκόλυνση τη διέλευση των συνόρων. Εδώ έχουμε το θέμα του RTP, του προγράμματος των εγγεγραμμένων ταξιδιωτών. Η πιο ελαφριά έκδοση του RTP που εξηγήθηκε στη μελέτη ως μια δεύτερη επιλογή και υπάρχει και η ιδέα του να μην έχουμε RTP αλλά να έχουμε ε, ουσιαστικά κάποια κέντρα επεξεργασίας και αυτό σχετίζεται με κάποια σχόλια που ακούσαμε από εσά ότι αυτή η συγκεκριμένη τρίτη επιλογή θα έπρεπε να συζητηθεί και εδώ, σε αυτό τον οίκο. Και φυσικά είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και μαζί σας. Να έχουμε και μια τεχνική συζήτηση όπως κάναμε και πέρσι για άλλα ζητήματα. Αλλά για αυτή την συγκεκριμένη υποεπιλογή των μελλοντικών προτάσεων που υπήρχαν στο χάρτη πορείας που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο μας ζητήθηκε να δώσουμε περαιτέρω εξηγήσει για αυτή την υποεπιλογή και το πράξαμε. Και είχαμε μια σύντομη συνεδρίαση και τότε προετοιμάσαμε και ένα ανεπίσημο έγγραφο, ένα paper, τον Αύγουστο που συζητήθηκε στην ομάδα Frontex με τα κράτη-μέλη. Και φυσικά σκοπεύουμε να έλθουμε και σε εσά να σας διαθέσουμε αυτό το έγγραφο για περαιτέρω συζήτηση. Όμως αυτό το έγγραφο είναι ένα non-paper και εξηγεί μία υποεπιλογή σε μία μελέτη εντυκτύπου που έχει δημοσιευθεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω όταν θα προετοιμάσουμε τις δικές μας προτάσεις αργότερα φέτος. Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο. Αφορά την περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων. Αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό θέμα που το διερευνούμε στη μελέτη δικτύπου και το πέμπτο μπλοκ ε, αφορά την πρόσβαση των διεκτικών αρχών, των αρχών επιβολής του νόμου σε αυτά τα δεδομένα. Αυτή είναι η ραχοκοκολιά ουσιαστικά της μελέτης αντικτύπου. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι η έναρξη της δημοσίας διαβούλευσης. Έγινε στις 29 Ιουλίου στην ιστοσελίδα της Κομισιόν και είναι ανοιχτή μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου για σχόλια, για feedback. Εμείς ε, ζητήσαμε από τις αντιπροσωπείες στο εξωτερικό να διαφημίσουν, ε, αν θέλετε, αυτή τη δημόσια διαβούλευση και έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει και οι κυβερνήσεις των τριτών χωρών να ενημερωθούν και θα έχουν και την ευκαιρία να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τίθεται στη διαβούλευση. Επίσης, ζητήσαμε και από την από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να απευθυνθεί στην κοινωνία των πολιτών, να συμμετέχουν οι πολίτες σε αυτή τη διαβούλευση και επίσης από την ίδια Λίσα ζητήθηκε να διαδώσει αυτή τη διαβούλευση και το αυτό θέλουμε να κάνουμε εδώ και σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή να γνωστοποιηθεί ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να απαντήσει κανείς λεπτομερώς στις ερωτήσεις που έχουμε θέσει. Και το τελευταίο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι είχαμε μια σειρά στοχευμένων συναντήσεων με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, τους ε, χάρη, τους αερομεταφορείς και τις ναυτιλικές εταιρείες, την κοινωνία των πολιτών, επίσης ε, με εκπροσώπους των διοικητικών αρχών, των αρχών επιβουλής του νόμου, με, των αρχών επιβουλής του με εκπροσώπους της ε, υπηρεσίας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και φυσικά τους επόμενους μήνες ε, έχουμε μία σειρά θεμάτων που θα συζητήσουμε στο πλαίσιο της μελέτης αντικτύπου. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν συνεχίζεται και θα πρέπει να έχουμε μία πλήρη αξιολόγηση για να υποστηρίξουμε αυτές τις πολύπλοκες προτάσεις που προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή. Και να επαναλάβω ότι όπως κάναμε και στο παρελθόν, σίγουρα θέλουμε να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις και μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Thank you for... Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Ο κύριος... Ε, Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Έχουν περάσει 70 ημέρες από τις 26 Ιουνίου και σήμερα από την πλευρά του κυρίου Ρόσενμπεργκ είδαμε ότι αναγνωρίστηκε η ύπαρξη αυτού του ανεπίσημου αυτού του non-paper. Θέλω να ενημερώσω την Κομισιόν την Επιτροπή, συγγνώμη, ο κ. Μωράες, εγώ και Τάνια γράψαμε μια επιστολή διαμαρτυρίας, έτσι όπως σας περιέγραψα πριν, με τους όρους αυτούς. Πάντως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο ότι όταν συνεδρίασε η ομάδα συνόρων στις 26 να είχαν ε, λάβει γνώση και οι συνεισηγητές για αυτό το ανεπίσημο έγγραφο και να θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί για αυτή την τρίτη επιλογή να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κέντρα και τους επιταχυντές που αναφέρατε. Πάντως σας ευχαριστώ και πάλι και ευχαριστώ και την υπηρεσία Γιουλής. Παρακαλώ. Εν συντομία, συμφωνώ με την άποψη ότι αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δίνονται σε ένα όργανο πρέπει και εμείς ενημερωνόμαστε. Συμφωνήθηκε με την Πρόεδρο να προσταθεί στην ημερήσια διάταξη μια επιστολή. Έχουμε συνάντηση συντονιστών, μάλιστα, δεν θα έχουμε ένα πρόβλημα. Άλλωστε, ε, έτσι μπορούμε όλε οι πολιτικέ ομάδε να συμφωνήσουμε να σταλεί αυτή η επιστολή το συντομότερο Δυνατών. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Κλείνουμε εδώ. Λίγο νωρίτερα από το πρόγραμμα αύριο μην ξεχάσετε τις κάρτες ψηφοφορίας, γιατί έχουμε ψηφοφορίες αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.